Welcome at Σας ε, καλωσορίζουμε σε αυτή την ε, συνεδρίαση. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αν δεν ε, έχει κανείς αντίρρηση για την ημερήσια διάταξη, νομίζω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε και νομίζω ότι έχουμε και πολύ καλά νέα σήμερα, γιατί μπορούμε να σας προσφέρουμε και τις 20 γλώσσες αυτό είναι το γλωσσικό προφίλ της συνεδρίασης. Το δεύτερο είναι ότι ε, να σας ενημερώσουμε για τους τριμερείς ε, διαλόγους, αλλά επειδή η κυρία Μπίσοφ δεν είναι εδώ, θα έρθει στις 10, θα το αναβάλουμε αυτό λιγάκι. Έγκριση των πρακτικών, αν δεν έχετε παρατηρήσεις ή κάποιες αντιρρήσεις, ε, νομίζω ότι μπορούμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Και έτσι λοιπόν ε, φτάνουμε στο θέμα της ε, ε, κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και αναγνώριση προσόντων στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Αυτή είναι μία μελέτη την οποία θα παρουσιάσει η κυρία Έλενα Φιρστές που είναι ερευνήτρια και η κυρία Ανταμισάσα που είναι project leader της εταιρείας Emilio Consulting. Δεν ξέρω αν είναι παρούσες οι κυρίες. Αν είναι παρούσες θα ήθελα να τις καλωσορίσω. Παρακαλώ λοιπόν, έχετε αν θέλετε το λόγο. Um, Good morning. My name is Elena tersch from Milieu. I'm here actually with my colleague Laura. Είμαι η ε, Έλενα και θα έρθει και η συνάδελφός μου και θα σας παρουσιάσουμε τη μελέτη μας για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και αναγνώριση προσόντων στα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Να σας ε, δώσω έτσι κάποιες ε, πληροφορίες όπως ε, ξέρετε, η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού βασίζεται στην ε, παροχή, ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως ακριβώς ε, προβλέπεται στην, στις συνθήκες και στην στρατηγική του 2020 για να υπάρχει καλύτερη, καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Νομίζω ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ ε, ανήκουμε ε, στο ενεργό δυναμικό 9,5 εκατομμύρια που μετακινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξ αυτών το 50% ε, βρίσκεται στη Γερμανία ή στην Αγγλία. Τα τελευταία 10 χρόνια οι εσωτερικές ροές αυξήθηκαν. Φτάσαμε περίπου στο 1 εκατομμύριο το 2017 οι χώρες προέλευσης της τελευταίας δεκαετίας ήταν Ρουμανία, Πολωνία και ακολουθούν Ιταλία, Πορτογαλία και Βουλγαρία. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ ή αργότερα στα βασικά κίνητρα γιατί εμφανίζεται αυτή η κινητικότητα. Αλλά η ανεργία είναι προφανώς ένα από τα βασικά κίνητρα. Ως εκ τούτου νομίζω ότι είναι καθοριστική σημασία οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να μπορούν να εργάζονται όταν μετακινούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος και να αναγνωρίζονται και τα προσόντα τους. Τώρα, όσον αφορά τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, αυτά στα διάφορα κράτη-μέλη ρυθμίζονται με διάφορους τρόπους. Το επίπεδο της ρύθμισης των επαγγελμάτων, τα είδη των επαγγελμάτων που ρυθμίζονται, η αυστηρότητα των ρυθμίσεων ε, ποικίλει στα διάφορα κράτη-μέλη σε γενικές γραμμές έχουμε περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ασκεί ε, επαγγέλματα που υπάγονται σε ρύθμιση, άρα δηλαδή αυτοί χρειάζονται κάποιο είδους ε, πιστοποίηση <clears throat> πριν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους. Και το σκεπτικό είναι να προστατεύονται, ε, προστατεύεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνολικός αριθμός ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπου 5.700 και οι τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ευστηρότητα είναι η υγεία, η ασφάλεια, η, δημόσιες, ε, η παροχή δημοσίων υπηρεσιών ε, Ω εκ τούτου τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει καταβάλει ε, πολλές προσπάθειες από τη δεκαετία του 60 για να προσφέρει αναγνώριση δεξιοτήτων σε άλλα κράτη-μέλη. Πριν λοιπόν ε, ρυθμιστεί αυτό το θέμα, το 2005 η οδηγία, εγκρίθηκε η οδηγία περί επαγγελματικών προσόντων και έτσι λοιπόν προέκυψε μια απλουστευμένη διαδικασία εναρμόνισης. Κατόπιν το 2011 υπήρξε αξιολόγηση αυτής της οδηγίας και αποκαλύφθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην αναγνώριση που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική πρόσβαση σε πληροφορίες και οι διαδικασίες είναι πολύ περίπλοκες. Έτσι λοιπόν η οδηγία αναθεωρήθηκε, η αναθεωρημένη οδηγία εγκρίθηκε το 2013. Τα κράτη-μέλη ήταν ε, υποχρεωμένα να εφαρμόσουν την οδηγία αυτή ε, στο εσωτερικό τους μέχρι το 2016. Τώρα λοιπόν η μελέτη μας ε, εξέτασε τις ε, αλλαγές σε αυτή την αναθεωρημένη οδηγία και εξέτασε αφενός ε, τα κενά και τους παράγοντες επιτυχίες ε, της ε, που προέκυψαν από την θεώρηση και από την άλλη προσπαθήσαμε να έχουμε μια πιο γενική γενική εξέταση των δεξιοτήτων το πώς αυτά σχετίζονται με άλλα εμπόδια στην κινητικότητα της εργασίας. Συνδυάζοντας αυτά, ε, θέλαμε να έχουμε μια καλύτερη γνώση ε, της ε, αναγνώρισης ε, προσόντων σχετικά με την κινητικότητα. Μελετήσαμε τα επαγγέλματα του τομέα υγείας, γιατί αυτό είναι ένας από τους τομείς όπου υπάρχουν πάρα πολλές ρυθμίσεις και είναι ένας καθοριστικός τομέας για τους μετακινούμενους εργαζόμενους. Κάναμε έρευνες, ανάλυση δεδομένων, συνεντεύξεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, κάναμε τέσσερις μελέτες περιπτώσεων και όλα αυτά για να μπορέσουμε να καλύψουμε μία σειρά χωρών, να καλύψουμε τις χώρες προορισμού, προέλευσης και διάφορα ρυθμιστικά μοντέλα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, τροποποίησεις, ε, ένα θέμα βασικό είναι η αμοιβαία αξιολόγηση και ο στόχος ήταν να αξιολογήσουμε κατά πόσον το είδος της αξιολόγησης εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για το στόχο μας και κατά πόσον θα μπορούσαν να αρθούν ε, κάποια εμπόδια. Αυτό λοιπόν κατέδειξε ότι η ποιότητα αξιολόγησης, ε, οι επιπτώσεις ε, ποικίλουν ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη ε, και δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές. Άρα δηλαδή δεν προέκυψαν σημαντικές αλλαγές στην προσέγγιση των κρατών μελών έναντι του κανονισμού. Και ως εκ τούτου το 2018 εγκρίθηκε μια οδηγία η οποία τώρα απαιτεί από τα κράτη-μέλη για οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση να εφαρμόζουν την αρχή της αναλογικότητας ε, για να μπορούν να αξιολογηθούν και οι κίνδυνοι από από μη ρύθμιση, στην περίπτωση δηλαδή που δεν προκύπτει ρύθμιση των επαγγελμάτων. Τώρα, ε, υπάρχουν και άλλες ε, τροπολογίες ε, στην έρευνα του 2013, όπου διαπιστώσαμε ότι αυτές οι αλλαγές έχουν σχέση με παροδική παροχή υπηρεσιών ή Διατάξει εκεί είναι λιγότερο αυστηρές. Μία άλλη αλλαγή αφορά την μερική ε, πρόσβαση. Έτσι λοιπόν μπορούν ε, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν ε, πληροφορίες για κάποια επαγγέλματα, αλλά όχι για όλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους δασκάλους των σχολείων. Σε γενικά όμως, σε γενικές γραμμές, αυτή η διάταξη δεν έτυχε και πολύ μεγάλης απήχησης. Κατόπιν, όσον αφορά στην εκπαίδευση. Τα κράτη-μέλη θεωρείται ότι θα μπορούσαν εθελοντικά να συμφωνήσουν σε θέματα εκπαίδευση για κάποια επαγγέλματα και έτσι να προκύπτει αυτόματα η αναγνώριση. Όμω στην περίπτωση αυτή ε, προέκυψε μόνο ένα πλαίσιο. Ε, μόνο εκεί μπορεί πλέον να γίνει αυτόματη αναγνώριση σε 11 κράτη-μέλη. άλλο, μια άλλη βασική αλλαγή του 2013 ήταν η επαγγελματική κάρτα που μπορεί κατ' ουσίαν να χρησιμοποιηθεί για έξι επαγγέλματα, μεταξύ αυτών ε, είναι και οι νοσοκόμες. Αλλά και αυτό ε, δεν χρησιμοποιήθηκε ικανοποιητικό, δηλαδή ανάμεσα στις νοσηλεύτριες μόνο το όσον ε, όσων ε, ζήτησαν την εφαρμογή αυτής της οδηγίας πέρασαν μέσα από τη ε, διαδικασία. Υπάρχουν λοιπόν, βλέπουμε, αρκετές διαφορές ανάμεσα στα επαγγέλματα και, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε περιορισμένη χρήση αυτής της δυνατότητας για αναγνώριση. Τα κράτη-μέλη εκλήθησαν να μελετήσουν ένα σημείο όπου οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ε, θα μπορούσαν να αποκτήσουν όλες τις ε, πληροφορίες για τη διαδικασία και αυτό θα έπρεπε να δώσει και τη δυνατότητα στους πολίτες να εφαρμόσουν ε, επιγραμμικά όλη τη διαδικασία της αναγνώρισης. Σε άλλα τέσσερα κράτη-μέλη όπου κάναμε σε βάθος μελέτες, ε, σε τρία κράτη-μέλη ήταν αδύνατον να υπάρξει περαιτέρω διαδικασία αναγνώρισης και στην Ολλανδία αυτό κατέστη τόν μόνο για κάποια επαγγέλματα. Εξάλλου, σε κάποια κράτη-μέλη υπήρχε έλλειψη πληροφοριών για τη διαδικασία και υπήρχαν και φραγμοί στη γλώσσα. Άρα δηλαδή η ενημέρωση προσφερόταν μόνο στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους, αλλά όχι σε άλλες δύο γλώσσες τουλάχιστον. Και υπάρχουν και κάποιες δύο άλλες αλλαγές ε, που δεν θα τις αναφέρω όμως, γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Σε γενικές γραμμές λοιπόν βλέπουμε ότι αυτές οι διατάξεις ε, και αυτές οι προϋποθέσεις ε, σε μεγάλο βαθμό ε, δεν χρησιμοποιήθηκαν. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω λιγάκι για τα βασικά αίτια της κινητικότητας και πώς ακριβώς παίζει ρόλο η αναγνώριση ή η μη αναγνώριση ε, στο να μπορεί κανείς να κινείται ευκολότερα ως εργαζόμενος. Όπως είπα και προηγουμένως, η απασχόληση είναι ένας ε, βασικός λόγος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί επιθυμούν να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος. Το 50% όσων ερωτήθηκαν είπαν ότι μετακινήθηκαν γιατί είχαν ήδη βρει μια άλλη θέση απασχόλησης ή ήθελαν να ε, βρουν κάποια άλλη θέση απασχόλησης. Μικρότερο είναι το ποσοστό που ανέφεραν οικογενειακούς λόγους, ε, εκεί συμπεριλαμβάνονται και οι σύζυγοι, ε, άρα δηλαδή εδώ έχουμε μία έμεση μετακίνηση. Η κινητικότητα για την απασχόληση ε, προκαλείται βέβαια από οικονομικούς και άλλους λόγους Κυρίως βλέπουμε διαφορές ε, στους ε, μισθούς, ε, στη διαβίωση, την μόνιμη εγκατάσταση. Αυτά τα βλέπουμε μετά την αύξηση της κινητικότητας το 2011 και το 2014, όταν δηλαδή ε, έπαυσαν να ισχύουν οι μεταβατικές ε, διατάξεις. Βλέπουμε αυξημένη κινητικότητα ε, ανάμεσα στις νοσηλεύτριες και στους, στο προσωπικό που παρέχει βοήθεια στο σπίτι. Διαπιστώνουμε την κινητικότητα ανάμεσα σε γειτνιάζουσες χώρες και κινητικότητα σε χώρες με την ίδια γλώσσα. Αυτά αφορούν και την ε, ε, διασυνοριακή κινητικότητα και μερικές φορές βλέπουμε ότι ο γλωσσικός παράγοντας υπερισχύει των διαφορών στους μισθούς. Ως εκ τούτου, η αναγνώριση ή η μη αναγνώριση είναι τελικά στοιχείο που διευκολύνει ή που εμποδίζει την κινητικότητα. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση, ούτε και έρχομαι και αρκετά δεδομένα, δεδομένα υψηλής ποιότητας για να μπορούμε να αποδείξουμε ακριβώς πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση σε σχέση με άλλους φραγμούς. Πάντως, εξετάζοντας τα θέματα της αναγνώρισης, βλέπετε είναι αυτή η πράσινη στήλη, διαπιστώνουμε ότι υπήρξε σημαντική αύξηση τα τελευταία 5 μέχρι 7 χρόνια. Και διαπιστώνουμε σε γενικές γραμμές ότι οι αποφάσεις περί αναγνώρισης ε, οδηγούν στο να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα, ε, θετικές αποφάσεις. Ε, αυτό είναι το 80% των αποφάσεων που λήφθησαν κατά την περίοδο που εξετάσαμε. Άρα δηλαδή η μη αναγνώριση καταλήγουμε στο ότι αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο σε αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν. Ε, βέβαια, στα στοιχεία που εξετάσαμε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν ε, σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα επαγγέλματα και στις ε, χώρες προέλευσης. Όσον αφορά τις χώρες προέλευσης, βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι οι νοσηλεύτριες από κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κροατία, αυτές έχουν θετική απόφαση γιατί σε αυτές παίζει ρόλο και το θέμα του μισθού. Ε, βέβαια έπρεπε να περάσουν μέσα από μία περίοδο προσαρμογής Ενώ όσον αφορά στις ε, νοσηλεύτριες από άλλες χώρες, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, το ποσοστό είναι σχεδόν μηδενικό. Και όσον αφορά τα διάφορα επαγγέλματα, βλέπουμε ότι υπάρχουν επαγγέλματα τα οποία εμπίπτουν σε συστήματα αριθμητικής αναγνώρισης, δηλαδή εκεί όπου η εκπαίδευση είναι εναρμονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αφορά τους γιατρούς και τις ε, νοσηλεύτριες. Ε, το ποσοστό των θετικών αποφάσεων είναι πολύ ψηλό, από 90 μέχρι 100%, Κατά τα άλλα ε, υπάρχουν επαγγέλματα που κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ε, το ποσοστό των θετικών αποφάσεων είναι λιγάκι χαμηλότερο, παραδείγματος χάρη για φυσιοθεραπευτές και για ε, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Εκεί το ποσοστό θετικής απόφασης κυμαίνεται από 60 μέχρι 80%. Επιπλέον, ε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτές οι τάσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την ομάδα των νοσηλευτριών. Αυτή είναι μια σημαντική ομάδα. Ε, η θετική απόφαση για αυτές είναι καθοριστική. Ε, περίπου το 1 τέταρτο των τάσεων είναι κατ' ουσίαν νοσηλεύτριες που ε, μετακινούνται σε ένα άλλο κράτος μέλος. Ε, για αυτές, αυτές ανέφεραν ότι η αναγνώριση των προσόντων τους σε άλλα κρατημέλη έπαιξε οπωσδήποτε ε, σημαντικό ρόλο. Αυτό αφορά κυρίως την αναγνώριση για τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Ρόλο έπαιξε η εναρμόνιση της εκπαίδευσης και το παράρτημα 5 της οδηγίας που επιτρέπει την αυτόματη αναγνώριση ορισμένων ε, τμήματων, κάποιας, κάποιων πτυχίων, κάποιας, ε, κάποιων τμήματων εκπαίδευσης. Φτάνοντας ε, λοιπόν στη σύγκριση αυτών των αριθμών, αν συγκρίνουμε το σύνολο των ροών, των μετακινήσεων, διαπιστώνουμε ότι τελικά λιγότερο από 10% είναι άτομα τα οποία μετακινούνται ε, χωρίς να έχουν ζητήσει την αναγνώριση. Αν το συγκρίνουμε αυτό με προηγούμενα ποσοστά, διαπιστώνουμε το 20% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εργάζονται σε ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ζητούν την αναγνώριση. Ε, βεβαίως ε, μπορούμε να ε, ρωτήσουμε και αν υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο ή αν ο μόνος παράγον που πειράζει είναι τελικά η αναγνώριση των προσόντων. απευθυνόμενοι στους Ευρωπαίους πολίτες διαπιστώνουμε ότι η έλλειψη ενημέρωσης και η μη αναγνώριση αποτελεί φραγμό στην κινητικότητα. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, το 4% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προσπάθησε να εργαστεί ή να σπουδάσει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αναγνώριση. τι οι άνθρωποι κατόρθωσαν να μετακινηθούν ε, και να εργαστούν ε, σε άλλη χώρα. Το ποσοστό τους είναι το ίδιο με άλλους που δεν κατόρθωσαν και από αυτό το 4% περίπου το 12% εξ αυτών ανέφεραν ότι η πρόσβαση στις ε, πληροφορίες ε, ήταν ένας φραγμός, ήταν ένα πρόβλημα για το ότι δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν σε άλλη χώρα. Και ένα άλλο 15% ανέφερε ότι η μη αναγνώριση από μελλοντικό εργοδότη ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα. Ως εκ τούτου η μη αναγνώριση είναι ένα θέμα που αφορά όχι μόνο την κινητικότητα, η μία αναγνώριση είναι και ένα εμπόδιο στο να βρει κανείς μια καλή δουλειά ανάλογα με τα προσόντα του. Όπως γνωρίζουμε, ε, το να έχει κανείς περισσότερα προσόντα από όσα ε, χρειάζονται. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά εκείνους που μετακινούνται και όχι τους υπόλοιπους. Ε, το 1 τρίτο όσων μετακινούνται ε, είπαν παραδείγματο χάρη ότι έχουν περισσότερα προσόντα από αυτά που χρειάζονται στη δουλειά τους. Αυτό αφορά ε, σε αυτούς που ε, παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας. Περίπου το 40% είπαν ότι έχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή ένα παρεμφερές πτυχίο. Άρα δηλαδή αυτοί δεν εργάζονται ανάλογα με τα προσόντα τους. Και όταν ρωτήσαμε το λόγο, πολλές φορές είπαν ότι είναι η γλώσσα, αλλά όχι μόνο αυτό, ε, σε κάποιες χώρες ε, υπάρχει και το πρόβλημα της μη αναγνώρισης των πτυχίων τους. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν ε, το τι μπορεί να γίνει και το τι μπορεί να βελτιωθεί, θέλω να πω, ε, θεωρώ ότι είναι απολύτως απαραίτητο να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες, το είδος των πληροφοριών για τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα και για τις διαδικασίες που ακολουθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πληροφορίες για την Τράπεζα Δεδομένων. Αυτό εξαρτάται βέβαια από το πόσο ξεκάθαρες είναι οι πληροφορίες στο κράτος μέλος. Ε, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι ιστοσελίδες. Ε, οι πρέπει να δίδονται και σε διάφορες γλώσσες. Ε, θα πρέπει να υπάρξει διαδικασία ευαισθητοποίησης για τα νέα εργαλεία, για την αναθεωρημένη οδηγία και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είπαν ότι είναι απαραίτητο να επικαιροποιείται το παράρτημα 5. Εκεί αναφέρονται ε, όλα τα μαθήματα αλλά και τα επαγγέλματα τα οποία είναι ρυθμιζόμενα. Εξάλλου υπάρχει ανάγκη και για περισσότερη έρευνα, δηλαδή να ε, συνεχιστούν αυτά που ξεκίνησαν με την, αμοιβέ, με την ε, διαδικασία αμοιβαίας αναγνώρισης, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της ρύθμισης των επαγγελμάτων. Και κατόπιν πρέπει να υπάρχει και ενδελεχής μελέτη των εμποδίων, ε, σχετικά με τις νέες ε, τροποποιημένες δυνατότητες που περιλαμβάνονται στην οδηγία. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε στοιχεία, πληροφορίες, μελέτες, ε, γιατί παραδείγματο χάρη οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν ανταποκρίθηκαν. Ως εκ τούτου πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω έρευνα σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σα ευχαριστούμε για την περίπλοκη, λέει η Πρόεδρος, αυτήν την παρουσίαση σχετικά με την κινητικότητα των κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Συνάδελφοι, μπορείτε τώρα να κάνετε τις ερωτήσεις. Οι συντονιστές θα ξεκινήσουν. Παρακαλώ. Έχουμε παρατηρήσει σχόλια επί του θέματος της παρουσίας αυτής. please. Um, Ο κύριος Πίσλαρο, ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα της μελέτης είναι αρκετά μέτρια ως νέα για μας. έως κακά ίσως είναι από τα πιο σημαντικά μέτρα που θα αύξαναν την ε, κινητικότητα και την αναγνώριση των επαγγελμάτων, το EPC, δεν χρησιμοποιείται σχεδόν. Δηλαδή, ίσως για τους οδηγούς των ορεινών διαδρομών είχε ένα αντίκτυπο, αλλά πραγματικά δείτε το αποτέλεσμα. Κάτω του 1% χρησιμοποιούν το εργαλείο αυτό που είχε αφιερωθεί στην υποστήριξη της επαγγελματική κινητικότητας. Το EPC σχετιζόταν και με την ψηφιοποίηση με του συστήματος ώστε να υπάρχουν κοινοποίησει ηλεκτρονικές μεταξύ των κρατών μελών. Δηλαδή, ως μέλος του Κοινοβουλίου ανησυχώ ιδιαίτερα. Εκπροσωπώντας τους πολίτες εδώ έχουμε σαφέστατα έλλειψη πολιτικής βούλησης σε επίπεδο κρατών μελών και έχουμε εμπόδια. Έχουμε εμπόδια εισόδου, εμπόδια κινητικότητες στην πραγματικότητα. Ήθελα λοιπόν ποιες, ποια, ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και ποιε θα ήταν οι πρακτικέ συστάσει που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε ώστε να βελτιώσουμε πραγματικά την κατάσταση. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Α ακούσουμε κάποια ερωτήματα και μετά τι απαντήσει. Η κυρία Ιουνκέρη, σε ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή που ήταν χρήσιμη Για μένα, στη δική μου χώρα, το να, μην δίνεται κανείς ε, από το Λίμπουργκ να εργαστεί στη Γερμανία στην ε, φροντίδα των μικρών παιδιών ή στο ένα ή το άλλο κομμάτι του Βελγίου είναι πάντα ένα πρόβλημα. Οι πολίτες μας ρωτούν γιατί δεν μπορείτε να επιλύσετε αυτή την κατάσταση να διευκολύνεται. Νομίζω λοιπόν ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα συμβαίνουν σε αυτήν ακριβώς την περιοχή των ε, κατοχυρωμένων ή ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων. Η πρόνοια, η φροντίδα των μικρών παιδιών, των ενηλίκων, των υπερηλίκων δηλαδή. Και η ερώτησή μου είναι τελείως αντίστοιχη με εκείνη του κυρίου Πισλέρου. Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι τα επόμενα μας βήματα. Πρέπει να ζητήσουμε αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Ή ε, μήπω δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό εμπόδιο. Μήπως χρειάζεται μια ενημερωτική εκστρατεία των κοινωνικών φορέων σχετικά με τα κατοχυρωμένα αυτά επαγγέλματα για να ερωτήσουμε κατά πόσον οι επίσημα απαιτητέ δεξιότητες είναι πράγματι αυτές που χρειάζονται. Γιατί έχουμε σημαντικές αποκλήσεις στις διάφορες χώρες. Στη Γερμανία θεωρείται ότι αν έχει 26 εβδομάδες είσαι καλυμμένος, στο Βέλγιο ή στην Ολλανδία 20 τέσσερις uh, Μήπως πρέπει δηλαδή να ηγηθούν τις προσπάθειες αυτής οι κοινωνικοί φορείς για το ποια ρύθμιση μας χρειάζεται. Madame Peter Hansen. Κυρία Πίτερ Χάνσεν, ευχαριστώ. Ε, ε, πρόεδρε για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Έχω πρώτα μία ερώτηση αντίστοιχη με εκείνη που έκαναν συνάδελφοι. Αν έχετε κάποιο παράδειγμα καλής πρακτικής από τα κράτη-μέλη, για να το δούμε. Και επίση τα ψηφιακά συστήματα, τι ρόλο έπαιξαν εδώ και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ίσως στο μέλλον. Η κυρία Ραφάλσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα είχα μία ερώτηση επί των θεμάτων έρευνας. Το πεδίο εφαρμογής για την έρευνα θα συνεχιστεί. Μάλλον η δική σας έρευνα ε, ε, περιορίστηκε σε κάποια μόνο κρατημέλη και σε, κάποιες, σε κάποιους μόνο τομείς, κυρίως εκείνο της πρόνοιας. Μπορείτε να αναλύσετε και άλλους τομείς όπως οι μεταφορές ή οι οικοδομές όπου υπάρχει υψηλότατη κινητικότητα μήπως έχουμε την ψευδέστηση ότι μπορούμε να προαγάγουμε την κινητικότητα μόνο μέσω νομοθετικής ρυθμίσεως. Γιατί τελικώς είναι μια προσωπική απόφαση επί τη βάση της κατάστασης στην αγορά απασχόλησης, επί τη βάση της ε, προσωπικής οικογενειακής κατάστασης του καθενός ή της γλωσσικής εγκύτητος προς κάποια άλλη χώρα ή περιφέρεια. Αλλά ναι, πρέπει να παρέχουμε το μέγιστο δυνατό αριθμό πληροφοριών. Θα πάμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων, ο κύριος Φούρλας. Κύριε Πρόεδρε, ε, σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα για ίση αμοιβή στην εργασία. Και δεν νομίζω να, πρέπει, να μπορούμε να είμαστε περήφανοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ξέρουμε ότι οι γυναίκε αμείβονται κατά 16% λιγότερο από του άντρε. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μέρα. Άκουσα με προσοχή ε, τα όσα αναφέρθηκαν, θα... πολύ απλή ερώτησή μου. Είναι απαραίτητο, λέει, να βελτιωθεί η πρόσβαση στις πληροφορίες. Ε, ανανέωση ιστοσελίδων, νέα εργαλεία. Πολύ απλό το ερώτημα. Ποιο θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ποιο θα μπει μπροστά για να τα υλοποιήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μποτέγκα, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εγώ διάβασα προσεκτικά την ε, μελέτη, την έκθεση αυτή. Ε, υπογραμμίζεται τον θετικό αντίκτυπο της ε, ρύθμισης επί των ε, μισθών των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσώτων. Ενώ αντίθετα λέτε ότι η έλλειψη ρύθμισης δεν εγγυάται τίποτα τέτοιο. Πιστεύω ότι είναι ένα συμπέρασμα σημαντικό και το ερώτημά μου εξ αυτού προέρχεται. Δηλαδή, η ανάπτυξη αυτού του μηχανισμού αναγνώρισης, του αυτόματου μηχανισμού αναγνώρισης. Μήπως θα έπρεπε να λαμβάνει υπόψη της και τον δυντικά αρνητικό αντίκτυπο επί των συνθήκων εργασίας ή άλλων συνθήκων στις χώρες όπου επιθυμούν να μετακινηθούν οι εργαζόμενοι. Μήπως θα έπρεπε να αποθαρρύνεται δηλαδή η ενίσχυση ε, σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς κατάρτισης ή μισθοδοσίας. Η κυρία Μπρουνέ, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για τη μελέτη αυτή. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Υφίσταται κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα Εράσμους για τα καταχειρωμένα αυτά επαγγελμάτα. Ιδιαίτερα για τα θέματα κατάρτισης. Γιατί ίσω αυτό θα μπορούσε πραγματικά να βελτιώσει την κατάσταση την κινητικότητα. Η κυρία Ροντιβέλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ερώτηση σχετικά με τα επαγγέλματα που εξετάζει αυτή η μελέτη. Ακούμε ότι οι διαδικασίες της αυτόματης αναγνώρισης που πρέπει να είναι το ελάχιστο κατόφλι αναγνώριση επαγγελματική, προποθέσει δηλαδή, περνούν από μια διαδικασία ή προσπάθεια εναρμόνιση ευρωπαϊκή και αυτή η αμοιβαία αναγνώριση των ελάχιστων προποθέσεων φαίνεται να λειτουργεί. Αλλά σε σχέση με την έρευνα που έγινε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει υψηλή κινητικότητα γεωγραφική και επαγγελματική στα επαγγέλματα που εξετάστηκαν εντό τη Ένωση. Επί τη βάση έρευνά σα, λοιπόν, πέραν της αναγνώρισης των ελαχίστων προσόντων. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια αναγνώριση ενωσιακή και του επίπεδου της επαγγελματικής δεξιότητας που με διαφορετικό τρόπο αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην φιλοξενούμενή μας για να απαντήσει ερωτήματα. Παρακαλώ. Thank you for the questions. For the first question... Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. περί των ε, εμποδίων για το EPC στη μελέτη μας έχουμε συμπεριλάβει κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελούν εμπόδια στη χρήση του EPC. Το ένα είναι πρακτική φύσεως, πρόκειται για την ενημέρωση, γιατί το EPC αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά γνωστό. Ένας λοιπόν από τους λόγους που δεν χρησιμοποιείται τόσο πολύ είναι αυτός. Έπειτα υπάρχουν δυσκολίες με την χρήση, πολύ με, τη χρήση του. Πολλοί αναφέραν δηλαδή ότι η χρήση του EPC είναι περίπλοκη. Ε, επίσης φαίνεται πως σε κάποια κράτη-μέλη προωθούν περισσότερο τη χρήση, ενώ άλλα όχι. Άρα λοιπόν μπορούν γι' αυτό να παρέμβουν οι αρχές των κρατών μελών. Διαφορετικά μπορεί και να οργανωθεί από, τα ευρωπαϊκά, από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς μια εκστρατεία ενημέρωσης για την ύπαρξη του EPC. Άλλο ζήτημα είναι, ε, ερώτηση μάλλον ήταν αν πρέπει να αναθεωρηθεί η ε, οδηγία ή αν χρειάζεται να υπάρξει περισσότερη ενημέρωση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά τόσο το Ευρωκοινοβούλιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι περισσότερο ζήτημα των κρατών μελών διότι πρόκειται για κανονισμό και ρυθμίσεις εντός των κρατών ε, μελών, α πούμε, διαφορά ανάμεσα στις Γερμανίδες ε, ε, νοσηλεύτριες και στις Ολλανδέζες νοσηλεύτριες όπου πληρώνονται περισσότερο γιατί η Γερμανία έχει αποφασίσει ότι αυτό το επάγγελμα ε, ε πρέπει να, έχει, να, να υπάγεται σε ψηλότερα πρότυπα. Δηλαδή ε, είναι θέμα των κατών μελών το αν θα αναρμονήσουν ή όχι τα προσόντα για συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ήδη υπάρχουν επαγγέλματα όπου είναι εναρμονισμένα και ρυθμισμένα τα προσόντα που πρέπει κανείς να έχει για επαγγελματική αναγνώριση, ε, γιατροί, αρχιτέκτονες ας πούμε, κάποια είδη νοσηλευτών, ε, Όπως σας είπα λοιπόν, είναι θέμα περισσότερο ε, κανονισμού. Ε, κρατών μελών. Η κυρία Φρίστερς, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός ο κανονισμός είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ μέσω της νομοθεσίας. Αυτό ωστόσο που είναι πολύ σημαντικό ε, δεν είναι η αναθεώρηση της οδηγίας και πάλι, αλλά η εξασφάλιση της σωστής μεταγραφής της. Το 2016 Υπήρξαν έλεγχοι ε, συμμόρφωσης που έγιναν για να ελεγχθεί η σωστή ε, μεταγραφή ε, και ξεκίνησαν διαδικασίες κατά παράβαση κατά σχεδόν όλων των κρατών μελών γιατί δεν είχε μεταγραφεί σωστά. Άρα λοιπόν πρέπει να ελεγχθεί ότι τώρα εφαρμόστηκε σωστά και ότι δεύτερον ότι, ότι έχει τεθεί και σε πράξη. Έπειτα, για τις ε, ψηφιακές ε, δεξιότητες. Ξέρουμε ότι το 40% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, που βεβαίως αν ε, θέλουμε να ψηφιοποιήσουμε το σύστημα αναγνώρισης, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό ο κόσμος, γιατί δεν έχει τις κατάλληλες δεξιότητες. Οπότε δεν θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Έπειτα, πρέπει να ενημερώσουμε και να κάνουμε την έρευνα Το θέμα είναι όμως ε, <coughs> ποιος διεξάγει την έρευνα, ποιος τη χρηματοδοτεί. Α πούμε, από πλευρά τη Κομισιόν έχει γίνει πολλή έρευνα για αυτό το θέμα, για την παιδεύση και τι ε, δεξιότητε, και αυτό φυσικά θα ε, συνεχιστεί. Ένα άλλο θέμα που ε, σχετίζεται με τις καλύτερες πρακτικές στα κρατη Για παράδειγμα, στη Γερμανία μπορούμε να δούμε ότι η Γερμανία έχει δημιουργήσει μια κεντρική αρχή για την αξιολόγηση ισοτήμων και αυτό καθιστά πολύ γρηγορότερη τη διαδικασία αναγνώρισης γιατί εν γέννη βεβαίως η αναγνώριση μπορεί να γίνει από διάφορα είδη αρχών, από επαγγελματικές ενώσεις, κάποιες φορές γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο, ας πούμε σε, ε, στη Γερμανία όπου οι περιφέρειες έχουν πολλές αρμοδιότητες, γίνεται εκεί σε αυτό το επίπεδο και έτσι είναι πολύ πιο εύκολο ε, γιατί είναι αποκεντρωμένη. Η αποκέντρωση λοιπόν αυτής της διαδικασίας και της αξιολόγησής της επιταχύνει συνήθως τη διαδικασία αναγνώρισης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Γερμανία και η Πολωνία που άρχισαν διάλογο και μάλιστα ανέπτυξαν κατάρτιση ε, στον τομέα της υγείας, ας πούμε κοινή κατάρτιση για τις νοσηλεύτριες με στόχο να διευκολυνθεί η κινητικότητα εργατικού δυναμικού ανάμεσα στις δύο χώρες. Με αυτόν τον τρόπο είναι πιο εύκολη η αξιολόγηση των προσόντων των επαγγελματικών του ίδιου τύπου σε δύο διαφορετικές χώρες. Ετέθη μια ερώτηση τώρα για το αν η αυτόματη αναγνώριση, η εναρμόνιση ε, έχει αρνητικό αντίκτυπο, για παράδειγμα, στις συνθήκες εργασίας. Πρώτα απ' όλα, δεν νομίζω πως η αναγνώριση αυτή η, ε, η εναρμόνιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε απορρίθμιση. γιατί υπάρχουν ε, οι ελάχιστες προδιαγραφές. Ας πούμε στην περίπτωση των ε, νοσηλευτών ε, θα αυξανόταν το επίπεδο δεξιοτήτων. Δηλαδή, Μπολόνια 3,2 ε, απαιτεί και πανεπιστημιακή κατάρτιση για τους νοσηλευτές. Ας πούμε, εναρμόνιση δεν θα έλεγα εγώ λοιπόν ότι θα οδηγήσει σε απορρίθμιση. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι για παράδειγμα έχει γίνει μελέτη για σύγκριση του αντικτύπου του κανονισμού στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και να δούμε κατά πόσο δηλαδή ε, υπάρχει ή όχι ε, πραγματικός αντίκτυπος. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο ο κανονισμός για κάθε επάγγελμα έχει αντίκτυπο στην πράξη. Αυτό θα πρέπει να γίνει λοιπόν σε επίπεδο κράτους μέλους ε, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε σωστά τον αντίκτυπο. Τώρα, θέματα που σχετίζονται με το, την οδηγία ε, έχουν να κάνουν με την επαγγελματική κατάρτιση μετά από την, ε, ε τις σπουδέ. Με το Erasmus Plus τώρα νομίζω μπορεί κανείς να κάνει και μαθητείες ε, και πρακτική εξάσκηση. Πάντως δεν είναι κάτι το οποίο καλύπτεται από την οδηγία. Και έπειτα ένα άλλο ζήτημα αφορά το κατά πόσο πρόκειται για ένα προσωπικό ζήτημα κατά το πόσο κινείται από ε, τις συνθήκες της αγοράς αυτό προσπάθησα να τονίσω, ότι η αναγνώριση ή μη δεν θεωρείται κίνητρο. Για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι από τη Ρουμανία είπαν ότι ο κόσμος δεν ε, μεταναστεύει επειδή τα προσόντα τους αναγνωρίζονται κάπου αλλού. Ε, το διευκολύνει αυτό βέβαια τη μετακίνηση, αλλά δεν είναι το βασικό ε, κίνητρο, όπως είναι ας πούμε η διαφορά στους μισθούς. Ξέρουμε ότι για κάποιες βασικές ε, θέσεις απασχόλησης στη Γερμανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή αυτές για τις οποίες χρειάζεται μόνο ε, πτυχίο, ε, απολυτήριο γυμνασίου, ξέρουμε ότι εκεί οι μισθοί στη Γερμανία και στην Βρετανία είναι ψηλότερες οι αποδοχές από ότι οι αποδοχές για κάποιες θέσεις με απαιτήσει ε, σπουδών στη Ρουμανία. Επίσης, ε, ο υπεριορισμός ε, και οι περικοπές στον τομέα της παιδείας αλλά και στον τομέα, στις αμοιβέ στις χώρες όπου επιβλήθηκαν μνημόνια είδαμε μεγάλη μετακίνηση πτυχιούχων από την Ιταλία και την Ισπανία και η Ιταλία δεν έχει ακόμα ανακτήσει όλες αυτές τις ροές και μάλιστα δεν έχουν αντιστραφεί οι ροές δηλαδή. Ακόμα υπάρχει μεγάλη ε, μετακίνηση Ιταλών. Φεύγουν από την Ιταλία δηλαδή. και είναι πιθανό ότι οι άνθρωποι θα μετακινηθούν ούτως ή άλλως, είτε αναγνωρίζονται δηλαδή τα πτυχία τους είτε όχι. Αλλά βέβαια, ειδικά εκεί όπου οι διαφορές δεν είναι και τόσο μεγάλες, οι διαφορές μισθών ή που έχουν ειδικά προσόντα, δεν θα μετακινηθούν εάν δεν αναγνωρίζεται η δουλειά τους, ή τα προσόντα τους, συγγνώμη, και δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά αλλού. Okay. I think that was it. Thank you. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε και όλα τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει στη συζήτηση αυτή και για τη συζήτηση μάλλον αυτή που είναι πολύ ενδιαφέροντα για μας. the Είναι πολύ χρήσιμα στοιχεία όσον αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων και σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα για να μας κάνετε την εισήγησή σας. Τώρα θα περάσουμε σε μια πολύ σύντομη ε, ψηφοφορία. It's not 10 o'clock yet, so we can either wait. Δεν είναι ακόμα 10 ακριβώς, είτε μπορούμε να περιμένουμε είτε να ξεκινήσουμε. Τι νομίζετε? Εντάξει, θα περιμένουμε. Μέχρι τις 10 ακριβώς, 4 λεπτά. Μετά θα ψηφίσουμε και μετά θα λάβουμε τις πληροφορίες ε, για τον τριμερή. It's 10 o'clock, my dear colleagues. So we will start with the vote. It's going to be a short one. Ε, λοιπόν, συνάδελφοι, πήγε 10 η ώρα, πρέπει να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ψηφίσουμε για το σχέδιο επιστολής ε, εκτιμώντας, εκτός από εκτιμώντας 3 και την παράγραφο 3. Ε, Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το εκτιμώντας 2 είναι πρόταση της Γκούε. Ποιοι είναι υπέρ. Ε, κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 3 πάλι πρόταση της γκουε, γκουε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική κλίση, οπότε παρακαλώ χρησιμοποιήστε τις κάρτες σας. Ready? Είστε έτοιμοι? Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία λοιπόν. Όχι κύριε Ουγγάριους. Ωραία. Τώρα τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, και τώρα πάμε στο σημείο 1, δηλαδή ενημέρωση για τον τριμερή για το AA3. Η κυρία Μπισχόφ έχει έρθει εγκαίρως. Οπότε μπορούμε να ακούσουμε την ενημέρωσή σας, κυρία Μπίσχοφ, που είστε και η συγγήτρια. Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους. Έχω καλά νέα να σας πω. Αν έχει την καλοσύνη να κάνετε ησυχία, γιατί ε, αυτά που θα ακούσουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, τα περιμένουμε όλοι εναγωνίως, <laughs> άρα να δώσουμε το λόγο στην ε, κυρία Μπίσοφ. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω το εξής. Ο ε, τριμερής διάλογος ε, για το 883 είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρξουν ε, πολλές αλλαγές στα κράτη-μέλη. Θα προσπαθήσουμε ε, για ένα θέμα που είναι πολύ περίπλοκο και στον ε, τριμερή διάλογο υπήρξαν αποτελέσματα, αλλά αυτά δεν εγκρίθηκαν στο Συμβούλιο. Είχαμε λοιπόν ήδη την πρώτη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου, όπου και οι δύο πλευρές ε, εξέφρασαν την προθυμία τους αυτή τη φορά να καταλήξουν σε συνένεση και να ολοκληρώσουν τις ε, διαπραγματεύσεις. Και επίσης, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι συντονιστές ε, συμφώνησαν ε, επί της εντολής και η CUP το στήριξε αυτό. Ε, Στιάσαμε την προσοχή μας ε, μόνο σε θέματα που είναι επίμαχα και δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στο Συμβούλιο. Και δεν θα ξεκινήσουν από την αρχή οι διαπραγματεύσει. γιατί αν το κάναμε αυτό, αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να τελειώσουμε. Ε, ε υπήρξε λοιπόν πάρα πολύ δουλειά, κατορθώσαμε να διαφυλάξουμε πάρα πολλά θέματα, περίπου το 80%, πάνω από 80% συμφωνήθηκε και στο 883 ξέρετε ότι αν όλοι είναι λίγο δυσαρεστημένοι αυτό είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ε, Εστιάσαμε την προσοχή μας σε θέματα επί των οποίων υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια ε, να σε ενημερώσω για το τι συμφωνήσαμε. Θα συζητήσουμε λοιπόν ε, για τα επιδόματα ανεργίας, για εργαζόμενους σε παραμεθόρειες περιοχές. Αυτό είναι ένα περίπλοκο θέμα, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις και στο Συμβούλιο και ως εκ τούτου περιμένουμε το Συμβούλιο να ε, μας δείξει συγκεκριμένα θέματα που θέλει να εξεταστούν και με τους σκιώδης ηγητές ε, θα προετοιμαστούμε πάρα πολύ καλά. Ε, θα περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει το Συμβούλιο και για τη δική μας τη στρατηγική. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το, το Κοινοβούλιο έκανε υποχωρήσεις, πολλούς συμβασμούς, αλλά πετύχαμε και πολλά πράγματα και θέλουμε να δούμε τελικά αν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συνένεση. Το δεύτερο σημαντικό είναι η νομοθεσία προς εφαρμογή. Ξέρετε ότι από αυτού υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις και εδώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ενημερώσω, θα ε, διαπραγματευτούμε επί του 85-86 και κάποιων άλλων ε, ρυθμίσεων και νομίζω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε ε, το τι επιτύχαμε στις τελευταίες διαπραγματεύσεις. Θα διαπραγματευτούμε τις διατάξεις 48, 71, 85, 86. Όπως σας είπα λοιπόν, στο Στρασβούργο θα έχουμε την Είχαμε την πρώτη συνάντηση του τρομερούς διαλόγου ανοιχτή συνάντηση, ορίσαμε τους στόχους και τώρα θα περάσουμε στην επόμενη φάση, στις, στην ουσία των διαπραγματεύσεων. Αλλά εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξη για το τελικό αποτέλεσμα. Είμαι ρεαλίστρια και γνωρίζω βέβαια ότι δεν μπορούν όλοι να είναι ικανοποιημένοι ε, με την τρέχουσα κατάσταση. Ως εκ τούτου και οι δύο πλευρές επιτιμούν να επιτύχουν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ κυρία Πίσοφ. Ε, να σας υπενθυμίσω ότι θα έχουμε δύο συναντήσεις. Η πρώτη είναι 7 Νοεμβρίου, η άλλη είναι 11 Νοεμβρίου πριν από τον επόμενο τριμερή διάλογο. Και επίσης ε, ε, στις 11 Νοεμβρίου θα έχουμε τον επόμενο διάλογο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πολύ καλά όλα αυτά που ακούσαμε. Εγώ θέλω το εξής, να μας πει η συγγήτρια αν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το θέμα του να ε, βελτιωθεί το επίδομα ανεργίας, ε, κατά πόσον αυτό ε, συζητείται στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου, γιατί ξέρετε αυτό συζητείται στα κράτη-μέλη εδώ και αρκετό καιρό. Η κυρία Μπίσοφ, μπορείτε να απαντήσετε, δεν ξέρω, θέλετε, επιθυμείτε να απαντήσετε ή μήπω δεν έχετε ακόμα την απάντηση σε αυτή την ερώτηση και ίσως μπορούμε αυτή την ε, ε, συζήτηση να την κάνουμε στο πλαίσιο των συντονιστών. Εν πάση αποφασίστε εσείς τι θέλετε να κάνετε. Καταρχήν θέλω να γνωρίζω αν έχετε και άλλες ερωτήσεις να τις κάνετε τώρα και να απαντήσω συλλογικά. Αν ε, δεν υπάρχουν άλλες, να απαντήσω τώρα. Αυτό τώρα δεν ήταν συζήτηση, ήταν περισσότερο ενημέρωση για τον τριμερή διάλογο. Η ε, κυρία Πίσοφ, κοιτάξτε, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο, αλλά πάντως ε, οι συντονιστές συμφώνησαν, ε, το Συμβούλιο συμφώνησε και θα περιμένουμε να δούμε. Ευχαριστούμε κύριος ε, Ράτκε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, λέει ο κύριος Ράτκε. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Κοιτάξτε, θα ήθελα να πω ε, Άκουσα από την ε, πρεσβεία μας ότι όσον αφορά τον τελικό στόχο ε, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Μπορεί λοιπόν κανείς να υποθέσει ότι αυτό το θέμα κατ' ουσίαν ε, έχει τεθεί εκτός συζήτηση ή μήπως ε, μπορεί κανείς να θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα έρχεται και θα επανέρχεται το θέμα έτσι ώστε να είναι και ένα αντικείμενο παζαριού για άλλα σημεία. Το Συμβούλιο συμφώνησε σχετικά με τον τελικό στόχο. Ήταν ε, πολύ ε, περίπλοκη όλη η συζήτηση, αλλά για το 883 τίποτα δεν είναι εύκολο. Ε, συμφώνησε λοιπόν το Συμβούλιο και η Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Και επίσης ε, και εγώ δεν θα ακολουθήσω αυτή τη γραμμή, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όσοι βρίσκονται σε αυτήν την αίθουσα. Αν ακολουθήσει κανείς αυτή τη γραμμή, έχει χάσει. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτύχουμε μια καλή συμφωνία. Και έχουμε δύο εκατομμύρια εργαζόμενους ε, στην Ευρώπη που περιμένουν να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και εμείς ε, παίρνουμε ενημέρωση, παίρνουμε πληροφορίες από το Συμβούλιο και θα δούμε τι θα γίνει στις 11 του μηνός όταν θα ξεκινήσει ο επόμενος ε, τριμερής διάλογος. Και μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό καλύτερα στην επόμενη συνεδρίαση των ε, σκιωδών και όλοι είμαστε, εν ε, σε επαφή και έχουμε και κάποιες πληροφορίες από το Συμβούλιο και θα δούμε πώς θα προχωρήσει το όλο θέμα. Κοιτάξτε, για μένα η διαφάνεια είναι καθοριστική σημασία ε, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και ως Κοινοβούλιο να παραμείνουμε ενωμένοι. Γι' αυτό είπα ότι ε, θα σας ενημερώσω μετά την πρώτη συνάντηση και θα συνεχίσω να σας ενημερώνω. Και αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ε, παρακαλώ, θα συνεχίσουμε να ερευνάμε την στρατηγική μας, να την καθορίζουμε τη στρατηγική μας και ε, να φροντίζουμε να είσαστε όλοι καλά ενημερωμένοι. Πολύ ωραία. Φτάνουμε τώρα σε μία παρουσίαση που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πρόκειται ε, για τους εργαζόμενους ε, που ε, εργάζονται στο θέμα στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Απασχόλησε το όμορφο με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. Πρόκειται για μια επιδημία και εξ όσων γνωρίζω, το ένα στα 10.000 παιδιά αυτό ήταν αναλογία το, κατά το παρελθόν αυτιστικό παιδί. Τώρα είναι το 1 στα 59 παιδιά που γεννιούνται. Το ένα στα 59 εντάσσεται στο αυτιστικό φάσμα. Οι αριθμοί όλο και αυξάνονται ο αριθμός των ανθρώπων που, που διαγνώσκονται ως άτομα με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος αυξάνεται όλο και περισσότερο ε, και οι περισσότεροι εξ αυτών παραμένουν άνεργοι. Ε, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα ε, όμως θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικοί εργαζόμενοι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε χρειαζόμαστε δεδομένα που θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, να βελτιώσουμε την ανταλλαγή ανάμεσα σε κράτη-μέλη, όπως επίσης και την ανταλλαγή επαγγελματιών σε όλους τους τομείς για να κατανοήσουμε καλύτερα τον αυτισμό. Η πιο σημαντική προϋπόθεση είναι ποιοτική έρευνα και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εδώ σήμερα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, θα ακούσουμε ακούσουμε την κυρία Αουρέλια Μπαράγκερ. Θα μας πείτε εσείς το όνομά σας με καλύτερη ε, προσφορά. Είναι Διευθύντρια του Οργανισμού Αυτισμού στην Ευρώπη. Θα μας παρουσιάσει την έρευνα των τελευταίων ετών, κυρίως όσον αφορά τις εξελίξεις στο θέμα της απασχόλησης ατόμων που εντάσσονται στο αυτιστικό φάσμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα μάλιστα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την ευκαιρία αυτή να σας παρουσιάσω ποια είναι η κατάσταση σχετικά με την απασχόληση των ανθρώπων με αυτισμό στην Ευρώπη. Όπως αναφέρατε υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού με διαταχές του αυτοιστικού φάσματος, περισσότερες διαγνώσεις και σήμερα θα αναφερθώ σε διάφορα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Καταρχά να θυμίσω λίγο για τα του αυτισμού και της απασχόλησης των ανθρώπων αυτών. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν για την πρόσβαση στην εργασία και ποια είναι και τα στοιχεία τα πιο θετικά ή τα πιο, ή πιο επιτυχημένες προσπάθειες. Έχουμε δει στο παρελθόν διάφορες πρωτοβουλίες ιδιαίτερα με τις νέες τεχνολογίες και σε αυτό θα αναφερθώ και μετά θα περάσω σε κάποιες συστάσεις για τους ηθήνοντες και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, να σας πω για την Autism Europe. Εμείς εκπροσωπούμε 90 ενώσεις και φορείς από 38 χώρες προσπαθώντας να υπερασπιστούμε των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αυτισμό με επικαιροποιημένε πληροφορίες και στοιχεία. Προάγουμε λοιπόν την έρευνα, προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τους ηθήνοντες πολιτικής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε μας υποστήριζε πολύ και επαναλαμβάνω με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα. Έχουμε πραγματοποιήσει πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωση μα έχετε υποστηρίξει και στο παρελθόν. Ελπίζουμε και φέτο να μα υποστηρίξετε γιατί θα έχουμε άλλη μια εκστρατεία επί των θεμάτων απασχόληση. Και πάμε ακριβώ στο θέμα για σήμερα. Καταρχά, σχετικά με τον αυτισμό. Ο αυτισμός χαρακτηρίζεται από δυσκολίες ε, στην κοινωνική επαφή και επικοινωνία και σύμφωνα με τα διαγνωστικά κριτήρια οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος έχουν συμπεριφορές επαναληπτικότητας υπερβολική ευαισθησία μερικές φορές στο φως στο ηλιακό φως που καθιστά πολύ δύσκολη την κοινωνική ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση. Χρειάζεται ειδικό φωτισμός για κάποιους από τους ανθρώπους αυτούς. Το συνολικό ποσοστό αποσχολησιμότητας των ανθρώπων με αυτισμό. Γνωρίζουμε ότι περί το 74% του γενικού πληθυσμού έχει απασχόληση. Αν πάμε στους ανθρώπους με αυτισμό πέφτουμε 48%. Μάλλον ανθρώπους με αναπηρίες είναι στο 48% για τους ανθρώπους με αυτισμό δεν έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία γνωρίζουμε ότι είναι πιο χαμηλό ακόμα το ποσοστό αυτό μία έρευνα που είχε διανεργηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέληγε ότι μόνο το 16% των ανθρώπων με αυτισμό είχαν πλήρη απασχόληση και 16% μερική απασχόληση. δεν έχει υπάρξει βελτίωση παρά τη βελτίωση του γενικού πληθυσμού ως προς την απασχόληση. Συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντως, έχουμε μια εκτίμηση ότι κάτω του 10% των ανθρώπων με αυτισμό έχουν θέση απασχόλησης, οι περισσότεροι σε προστατευμένες συνθήκες και σε θέσεις απασχόλησης χαμηλής αμοιβή. οι περισσότεροι από αυτούς που λαμβάνουν μια υποστήριξη δεν συμπεριλαμβάνονται αναγκαστικά στα στατιστικά στοιχεία και συνήθως λαμβάνουν πολύ περισσότερη υποστήριξη από τον οικογενειακό τους περίγυρο. Η έρευνα επίσης μας έχει δείξει ότι ακόμα και αυτοί που έχουν δεξιότητες ή προσόντα υψηλότερες του μέσου όρου τείνουν να έχουν μια θέση απασχόλησης χαμηλής αμοιβή, χαμηλού μισθού και πάντως χαμηλότερου από αυτού που θα δικαιολογούσαν οι δεξιότητές τους. Έχουμε εμπόδια που σχετίζονται με τον αυτισμό, δυσκολίες επικοινωνίας, θα δούμε και ένα βίντεο που θα μας εξηγεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί όταν καλούνται να έχουν μια συνέντευξη για πρόσληψη. Υφίστανται διάφορες διακρίσεις και στην πρόσβαση στην παιδεία. Έχουν ψηλά ποσοστά εγκατάλειψης των σχολικών και άλλων σπουδών, διότι δεν μπορούν να λάβουν την πλήρη υποστήριξη που χρειάζονται. Έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην επαγγελματική κατάρτιση και υπάρχουν και διάφορες προκαταλήψεις μεταξύ του πληθυσμού. Υπάρχει μια ανισχία ή ένας φόβος, αν θέλετε, καχυποψία πλευράς των εργοδοτών. Μια έλλειψη εμπιστοσύνη στις δεξιότητες και τις ικανότητες των ανθρώπων με αυτισμό και υπάρχουν εμπόδια και στην διαδικασία της πιθανής πρόσληψης. Θα δούμε ένα σύντομο βίντεο τώρα που προετοίμασαν τα μέλη μας από τη Βρετανία και που δείχνουν τις δυσκολίες προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί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 unemployable. I'm autistic, and sometimes I get too much information. So this video illustrates... Αυτό το βίντεο λοιπόν δείχνει πολύ καλά κάποια από τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αυτισμό με έλλειψη καταλήλων χώρων για τις συνεντεύξεις τους, ε, με έλλειψη πιο συγκεκριμένων ερωτημάτων που θα πρέπει να τους απευθύνονται ή περισσότερου χρόνου που θα έπρεπε να έχουν στην διάθεσή τους, όπως είδατε. Είχαμε μια άλλη έρευνα στο Ηνωμένο Βασίλειο που μας δείχνει ότι το 42% των ε, ενηλίκων με αυτισμό θα, χρειάζονταν υποστήριξη απασχόλησης μόνο το 12% το λαμβάνει. Το 13% λέγει ότι κάποια από την υποστήριξη τους βοηθάει στην αναζήτηση θέσης απασχόλησης, αλλά το 37% λέει, ε, λέει ότι θα χρειαζόταν πολύ περισσότερη υποστήριξη ενώ μόνο το 4% λέει ότι το προσωπικό που ασχολείται μαζί τους, που επικοινωνεί μαζί τους, έχει τις κατάλληλες ικανότητες για να το κάνει. Νομίζω όμως ότι πρέπει να αναφερθούμε και στα θετικά στοιχεία, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχει δυναμικό, γιατί ναι υπάρχουν εμπόδια, αλλά υπάρχει και μια και η άλλη όψη του νομίσματος, οι έρευνε μας έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι με αυτισμό είναι πάρα πολύ καλοί στην συστηματοποίηση. Είναι πολύ καλοί στην ε, οπτικοποιημένη σκέψη και έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σε συγκεκριμένες θεματικές. Είναι πολύ μεθοδικοί συνήθως είναι πολύ παρατηρητικοί και σκέπτονται με διαφορετικό τρόπο. Επομένως έχουν νέες προσεγγίσεις, καινοτόμες προσεγγίσεις για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι σε θέση να συνεισφέρουν σημαντικά με δημιουργικό τρόπο στην επιστημονική έρευνα. Επίσης είναι απολύτως ειλικρινής και αξιόπιστη Βεβαίω ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη. Είναι σημαντικό να οικοδομήσει, πιστεύω κανείς, επί των θετικών αυτών στοιχείων ώστε να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα απασχόλησης. Κάποιες από τις αρχές λοιπόν τα πορίσματα της έρευνας που έχει γίνει είναι ότι προκειμένου να έχουμε μια αποτελεσματική υποστήριξη απασχόλησης πρέπει να εστιαστούμε στις, στα πιο θετικά στοιχεία, στα πλεονεκτήματα των ανθρώπων με αυτισμό πρέπει να περιγράψουμε και να αντιληφθούμε καλύτερα τις ανάγκες τους αλλά και τις ιδιαιτερότητες τους χρειάζονται ε, χώρο με προστασία από το θόρυβο και κυρίως το φως και είναι σημαντικό να υπάρχουν κάποια προγράμματα επαγγελματικής εμπειρίας ώστε να μαθαίνουν και επί το έργο. Οι εργοδότες χρειάζονται καλύτερα ποσοτικά στοιχεία, χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση σε πόρους, σε κονδύλια για την ενίσχυση και προστασία των ανθρώπων με αυτισμό και βεβαίως οι εργοδότες έχουν μια ευθύνη να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση, επίγνωση της παρουσίας του προβλήματος αυτού στο χώρο της εργασίας. Σορεύονται τα εμπόδια ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίε και είναι σημαντικό να γίνει μια δουλειά και στον τομέα της παιδείας ενημερωτικά. Πάντως μπορούν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί εφόσον έχουν την κατάλληλη υποστήριξη και το κατάλληλο πλαίσιο για τη δουλειά τους. Οι άνθρωποι με αυτισμό. Έχουμε παραδείγματα από τις νέες τεχνολογίες. Επίσης μπορεί να προσαρμοστεί το προφίλ μιας συγκεκριμένης θέσης απασχόλησης προς τις δεξιότητες ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Αλλά ε, σημειώνονται κενά ευκαιρίας και τελικώς σημαντική δυσκολία στις προσλήψεις ανθρώπων με αυτισμό. Υπάρχουν όμως και αναγνωρισμένα δικαιώματα υπό τα Ηνωμένα Έθνη για τους ανθρώπους με αναπηρία σε μια προστατευμένη θέση απασχόλησης εφόσον προσπαθούμε να προωθήσουμε την γνώση κύκλου ζωής ε, και τις ε, επαγγελματικές δεξιότητες με προγράμματα κατάρτισης μπορούμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των ανθρώπων με αυτισμό αλλά θα έπρεπε να στοχεύουμε στην, στην ανοιχτή αγορά απασχόλησης. Πάντω είναι σημαντικό να υπάρχει εξειδικευμένη καθοδήγηση και παροχή συμβουλών. και πριν την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της απασχόλησης. Είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει ένα, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για τις συνεντεύξεις πρόσληψης, για τις ερωτήσεις που θα απευθύνονται στους ανθρώπους με αυτισμό και να υπάρχει μια επίγνωση των εργοδοτών και των συναδέλφων καθ' όλη τη διάρκεια της απασχόλησης. Έχουν αναπτυχθεί κάποια προγράμματα ιδιαίτερα στην τεχνολογία της πληροφορίας υπάρχει το Specialistern στη Δανία, το οποίο εκκίνησε προκειμένου να δημιουργήσει ένα εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης για ανθρώπους με αυτισμό, σε συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις, με πέντε μήνες πρόγραμμα κατάρτισης για κάθε άνθρωπο με αυτισμό που συμμετείχε, και υπάρχουν αρκετέ εταιρείε που έχουν συσχετιστεί με το πρόγραμμα αυτό. Το Passwerk στο Βέλγιο, η Oticon στη Γερμανία, πρόκειται δηλαδή για πρότυπα που λειτουργούν προκειμένου να παράσχουν υποστήριξη για καθοδήγηση στον χώρο εργασίας αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι οι άνθρωποι με αυτισμό στις νέες τεχνολογίες ή στην ψηφιακή τεχνολογία. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν τα πράγματα αυτά σε διάφορους τομείς. Άλλες έρευνες μας έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι με αυτισμό έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τέχνες ή τα διοικητικά επαγγέλματα τύπου επαγγελμάτων στη βιβλιοθήκη για παράδειγμα. Ε, με κάποια επαγγέλματα ή κάποια θέση που να έχει μια οργανωτική διάσταση ή διαχειριστική διάσταση. Και πάω στο τελευταίο τμήμα της παρασίασής μου για να θυμίσω λίγο το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχουμε σε ενωσιακό επίπεδο. Θα γνωρίζετε ότι όλα τα κρατημέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επικυρώσει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, το άρθρο 27 για την απασχόληση, για την πρόσβαση στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Επανεξετάζοντας λοιπόν την υλοποίηση της σύμβασης το 2015, η Επιτροπή CRPD ετώνησε ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν μέτρα καλύτερης γνώσης του ποσοστού απασχόλησης των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε να αυξηθεί η απασχολησιμότητά τους, ιδιαίτερα για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ε, ψυχοκοινωνικές ε, αναπηρίες ή δυσκολίες. Δηλαδή αυτό που συζητούμε. Επίσης υπάρχει ο στόχος υπαριθμών 8 για την υποστήριξη των ανθρώπων με αναπηρίες, Υπάρχει και η οδηγία ισότητα στην εργασία για την ε, εξάλληψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των Κοινωνικών Δικαιωμάτων για την ε, ενεργό στήριξη προ την απασχόληση και για την παροχή υπηρεσιών ώστε να υποστηρίζονται οι άνθρωποι με αναπηρία στην αγορά εργασία. Έχουμε δηλαδή ένα πλαίσιο εντό του οποίου μπορούμε να εργαστούμε ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και έχουμε και κάποιες συστάσεις για τους εθνικούς ηθήνοντες, αλλά και για το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συλλογή των στοιχείων είναι πάρα πολύ σημαντική έχουμε λίγα στατιστικά στοιχεία για τους πραγματικούς αριθμούς ανθρώπων με αυτισμό που απασχολούνται σήμερα και είναι σημαντικό να θέσουμε στόχους ώστε να βελτιώσουμε την απασχόλησή τους χρειάζονται εξειδικευμένες υπηρεσίες στήριξης σε όλη τη διάρκεια της απασχόλησης και πρέπει να προωθήσουμε το δυναμικό, τις δυνατότητες που έχουν οι άνθρωποι αυτοί για τους εργοδότες συνολικά. Είναι σημαντικό επίσης να επενδύσουμε στην ερευνά ώστε να παρακολουθούμε και τα αποτελέσματα και να αναπτύξουμε πιο αποτελεσματικά προγράμματα επίσης να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι υπηρεσίες από ανθρώπους που θα έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση, κατάρτιση, ώστε να επικοινωνούν με ανθρώπους με αναπηρίες και κυρίως ανθρώπους με αυτισμό, να έχουμε πιλωτικά προγράμματα κατάρτισης για να δούμε τι λειτουργεί καλύτερα και ιδιαίτερα στη, στη δημόσια διοίκηση θα πρέπει να υπάρξει ένα παράδειγμα για το υπόλοιπο της αγοράς απασχόλησης ώστε να καλυφθεί η παγίδα των επιδομάτων. Δηλαδή συχνά υπάρχει μια, ένας, μια διστακτικότητα να περάσει κανείς στην αγορά απασχόλησης εγκαταλείποντας το επίδομα που ενδεχομένως λαμβάνει. Για το ευρωπαϊκό επίπεδο πιστεύουμε ότι πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια ισχυρή και φιλόδοξη στρατηγική για τις αναπηρίες για την περίοδο 2020-30. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από επαρκείς πόρους και θα πρέπει να διοχετευτεί σε όλες τους τομείς πολιτικής συμπεριλαμβανομένης της εργασίας. Αυτό δεν μπορεί παρά να απαιτεί έναν ισχυρό μηχανισμό συντονισμού που είναι μια προσδοκία για τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να προτείνει μια νέα οδηγία επίσης ώστε να έχουμε μια εναρμονισμένη κατανόηση σχετικά με τις υποδημές που χρειάζονται για τους ανθρώπους με αυτισμό. Επίσης είναι σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βελτιώσουμε την συλλογή των δεδομένων ανά είδος αναπηρίας και ελπίζουμε να υπάρξει ένας ισχυρός κανονισμός για το ESF Plus, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ειδικά για τους ανθρώπους με αναπηρία και υπάρχει και η ελευθερία μετακίνησης και εργασίας στο εξωτερικό και για τους ανθρώπους που έχουν διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Ενώ αυτή τη στιγμή αναγκάζονται να περάσουν από διάφορες διαδικασίες αξιολόγησης. Και αυτές οι αξιολογήσεις χρειάζονται εναρμόνιση, Χρειάζεται να υποστηριχθεί η έρευνα και οι κοινωνικές επενδύσεις για πρωτοβουλίες κοινωνικής συμπερίληψης και ένταξης και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηγετικό ρόλο και ευθύνη στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που θα πρέπει να γίνεται βεβαίως με τις οργανώσεις, τις ενώσεις, τους φορείς που εκπροσωπούν τους ανθρώπους αυτούς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη όσον αφορά το ναυτισμό και τις σχετικές πολιτικές. Υπάρχουν χώρες όπου κάνουν φοβερά πράγματα όπως η Πολωνία και μετά, ε, όπως η Νορβηγία με συγχωρείτε και έπειτα υπάρχουν χώρες όπως η Σλοβακία πράγμα για το οποίο ντρέπομαι φρικτά που κάνουν ελάχιστα πράγματα διοργανώσαμε μια διάσκεψη στη Σλοβακία για τα αυτιστικά του αυτιστικά άτομα και τα αυτιστικά παιδιά και με μεγάλη θλίψη άκουσα τα γεγονότα, τα στοιχεία, τις ιστορίες που άκουσα εκεί. Δηλαδή, όχι μόνο ότι αποκλείονται από το ναι, εκπαίδευση αλλά και από την αγορά εργασίας και από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Οι κύριοι μας προσκεκλημένοι ήταν άνθρωποι από την κοινωνία με το σύνδρομο Άσπεργκερ, πολύ συχνά με μεγάλο επίπεδο, ψηλό επίπεδο IQ, αλλά πολύ χαμηλό επίπεδο κοινωνικών δεξιοτήτων. Με μεγάλη θλίψη λοιπόν άκουσα τις ιστορίες τους, γιατί συνήθως είναι πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, έχουν πτυχία πανεπιστημιακά και είναι σε θέση να συμβάλλουν στην κοινωνία ακόμα και αν το επιθυμούν λοιπόν βαθιά, η κοινωνία διαρκώς τους ε, απαρνείται. Πολύ δύσκολο, μεγάλος αριθμός ε, αυτών των ανθρώπων σε νέα ηλικία ε, αυτοκτονούν, ακριβώς επειδή κατά σύστημα η κοινωνία τους απαρνείται. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ λυπηρό. Και ειλικρινά πιστεύω πως κάτι θα πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για τις συστάσεις που μας κάνετε και τώρα θα λάβετε το λόγο ε, από την Επιτροπή ε, όποιος θέλει. Πρώτη η κυρία Κόφη. Η κυρία Μπρόφη, σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την εξαιρετική σας ε, ε, εισήγηση. Η ερώτησή μου αφορά το 1% του πληθυσμού της Ένωσης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι μόνο 16% των ανθρώπων με αυτισμό γνωρίζουν ε, τις πολιτικές που υπάρχουν. Πολύ χαμηλό το ποσοστό και είναι ιδιαίτερα λυπηρό γιατί όπως είπατε περισσότερα οι, οι ε, αυτιστικοί άνθρωποι έχουν πολύ ψηλό IQ και ε, μόρφωση. Η, Δυστυχώς ε, οι άνθρωποι με αυτισμό δεν εκτιμούνται από τους χώρους εργασίας και μάλιστα η έκθεσή σας δείχνει και ότι κάποιοι άνθρωποι δεν, αυτιστικοί δεν παρακολουθούν ε, ε, κάποια εκπαιδευτικά ε, προγράμματα. Νομίζω πως μπορούμε λοιπόν να κάνουμε περισσότερα πράγματα και θα, θα σας πω κάτι προσωπικό γιατί έχω έναν 26χρονο γιο που ε, πάσχει από αυτισμό. Αγωνίστηκε στα, σχολικά χρόνια, είναι εξαιρετικά έξυπνος, έχει πετύχει τον ψηλότερο δυνατό βαθμό στα μαθηματικά και κατάφερε να φτάσει στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς λόγω της έλλειψης υποστήριξης για την εκείνον ε, ε, στα σχολικά του χρόνια δεν μπόρεσε να προχωρήσει πέρα από το δεύτερο έτος γιατί είχε καταστροφικά αποτελέσματα λόγω ψυχικών προβλημάτων <coughs> που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν. Πολλοί αυτιστικοί άνθρωποι το παθαίνουν αυτό. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι στα κρίσιμα αυτά χρόνια ανάπτυξης όλοι οι άνθρωποι που υποφέρουν από αυτισμό, ειδικά αυτοί που έχουν τόσο μεγάλο ταλέντο, να μην μένουν εκτός του συστήματος Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την ψυχική υγεία των νέων ε, που πάσχουν από αυτισμό. Πιστεύω πως ε, θα πρέπει να προστατεύονται τα παιδιά αυτά σε αυτά τα τόσο κρίσιμα χρόνια ε, στην νεαρή του ηλικία δηλαδή. Η ψυχική υγεία θα πρέπει να προβλέπεται, να προσφέρεται στη διάρκεια των, των χρόνων όπου τα παιδιά αυτά παρακολουθούν το εκπαιδευτικό ε, σύστημα. Πώς μπορούμε να το στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, πραγματικά εξαιρετική ομιλία. Νομίζω ότι σε ορισμένα ε, θέματα καταστήσατε απόλυτα σαφές ότι οι άνθρωποι με αυτισμό είναι συγκεκριμένες προσωπικότητες και δεν μπορεί κανείς να πει ότι πρέπει στις περιπτώσεις αυτές ε, να γίνει το α ή το β. Δεν υπάρχει κάτι το ε, συγκεκριμένο ε, και γι' αυτό λοιπόν εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν μ' αρέσει ο όρος πόνος και συμπόνια. Ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς, ε, γιατί ε, για τα άτομα με αυτισμό αυτό δεν ισχύει. Ε, τα άτομα με αυτισμό πιστεύουν ότι ο υπόλοιπο κόσμος δεν ταιριάζει σε αυτούς. Και ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή προσέγγισης. Δηλαδή να καταλάβει η κοινωνία ότι τα παιδιά με αυτισμό αισθάνονται θαυμάσια, απλά πιστεύουν ότι οι υπόλοιποι έχουν κάποιο πρόβλημα. Εξάλλου πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα άτομα με αυτισμό ε, προφανώς έχουν δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αυτό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Δεν είναι θέμα καλής θέλησης. Η σα έθιξε το θέμα της ε, εκπαίδευσης. Βεβαίως και τα νέα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση και ούτως ή άλλως και στην περίπτωσή τους ισχύει η αρχή περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων η εργασία πρέπει να προσαρμόζεται στον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος στην εργασία σε αυτή την ειδική περίπτωση. Κατά τη δική σας άποψη, τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να επιτύχουμε βελτιώσεις. Τι θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να έχουμε παραδείγματα βέλτιστων ε, πρακτικών ε, πού ε, πρέπει κανείς να στρέψει την προσοχή του, τι μπορούμε να στηρίξουμε. Όπως είπε και η Πρόεδρος, ε, στην Νορβηγία τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ε, σε άλλες χώρες υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Μπορείτε να μας ενημερώσετε λίγο καλύτερα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κιμπουρόπουλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά η εισήγηση ήταν μια πολύ ωραία εισήγηση που ε, περιγράφει, θα πω, όχι μόνο για τους αυτιστικούς συμπολίτε μας μια αληθινή κατάσταση, αλλά μια, ε, για όλους τους ε, ανάπηρους συμπολίτε το τι συμβαίνει στην, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, η αλήθεια είναι ότι μέσα στην εισήγηση αναπτύχθηκαν πολλά θέματα ε, επιδόματα, προστατευόμενη εργασία, ε, μεγάλο ποσοστό φτώχειας, ε, ανεργίας συγγνώμη, και φτώχειας στους αυτιστικούς συμπολίτες μας. Εγώ έχω μία ερώτηση προς την εισηγήτρια και μία πρόταση ε, επίσης. Όλα αυτά βέβαια τα θέματα που του την πρόταση και την ερώτηση είναι Αυτά τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν από την εισηγήτρια πρέπει και χρειάζεται εδώ στην Επιτροπή μας να τα δούμε και να τα αξιολογήσουμε για περαιτέρω συζήτηση. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς ο οργανισμός σας και αν ε, συνεργάζεται με άλλους ε, οργανισμούς που ασχολούνται με την αναπηρία για να λύσουν αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι θέματα που αφορούν μόνο τον αυτισμό, αλλά αφορούν συνολικά την αναπηρία. Και δεύτερον, θεωρώ ότι οι εταιρείε πρέπει να δέχονται μια εκπαίδευση για το πώς θα συμπεριφέρονται σε ανάπηρους συμπολίτε μας. Πρέπει να δέχονται μια επιπλέον ε, εκπαίδευση για τις ερωτήσεις, για τον τρόπο που παίρνουμε συνεντεύξεις, γιατί δεν είναι μόνο ο αυτισμό που δέχεται αποκλεισμό, αλλά είναι και οι υπόλοιπε αναπηρίε. Και αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά σε ολόκληρο το επίπεδο τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Mr. please. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Η συζήτηση που κάναμε δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Η πρόεδρος ε, επισήμανε ε, το ποιε θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις ε, στις διάφορες χώρες. Θέλω να σας πω ότι και στη δική μου τη χώρα, την Πολωνία, τα πράγματα δεν είναι εξαιρετικά, αν και τα τελευταία χρόνια πρέπει να πω ότι έχει σημειωθεί μια κάποια πρόοδος. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε, νιώθουμε φόβο. Ε, φοβούμεθα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένοι σε μια εύρυθμα λειτουργούσα κοινωνία. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και πρέπει να, πρέπει, θέλω να καλέσω όλους να ε, αλλάξουν μέσα από την ευαισθητοποίηση την νοοτροπία των ανθρώπων. Γιατί οι φραγμοί βρίσκονται σε εμά, μέσα στο δικό μας τον εγκέφαλο. Ε, θέλω λοιπόν να αναφερθώ λιγάκι και σε θέματα εργασίας ανθρώπων με αυτισμό. Νομίζω το σημαντικότερο όλων είναι η εκπαίδευση. Τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι το 26% των ατόμων με αυτισμό εργάζονται. 72% ε, είναι τα ποσοστά των ατόμων με αυτισμό που έχουν πτυχίο πανεπιστημίου και εργάζονται. Άρα δηλαδή βλέπετε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της εκπαίδευσης. Υπάρχουν βέβαια και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις που πρέπει να στηριχθούν. Ένα τέτοιο πολύ καλό ε, παράδειγμα, κατά την άποψή μου, είναι το Autista at Work. Πολύ καλό παράδειγμα αυτό και θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα παρεμφερή παραδείγματα. Ως εκ τούτου, το βασικό ερώτημα είναι το τι πρέπει να γίνει πώς να στηρίζεται η απασχόληση, ε, κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, σύμβουλος ε, και νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχουν και βοηθητικά εργαλεία. Στην παρουσίαση ετέθησαν και κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τη δική μου τη χώρα, δηλαδή Στη δική μου τη χώρα υπάρχει δυστυχώς η παγίδα της απόδοσης και αυτή η παγίδα αποκλείει άτομα με αυτισμό από την αγορά εργασίας. Θέλω λοιπόν να ερωτήσω, ε, η Autist Europe, ο οργανισμός αυτός, έχει να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Γιατί στη δική μου τη χώρα υπάρχει το πρόβλημα ότι πάρα πολλοί πέφτουν σε αυτή την παγίδα της απόδοσης και είναι πολύ δύσκολο να βγουν από αυτήν. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια γιατί το θέμα είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Ντούρα Φερνάντε, παρακαλώ. Ντούρα Φερνάντης, ε, πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα μιλήσω στα ισπανικά. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μας διαβάζει μια εικόνα όχι μόνο των δυσκολιών και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αυτισμό, αλλά και των δυνατοτήτων τους. Γιατί πιο συχνά εστιαζόμαστε στα προβλήματα, παρά στις δυνατότητες που θα μπορούσαμε να έχουμε. Υποτένει αυτή μου άρεσε πολύ η παρουσίαση και ίσως θα έπρεπε ανάλογα με το δυναμικό του καθενός να έχουμε μια προσπάθεια καλύτερης ένταξης. Όπως υπόθηκε υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς την εργασιακή ένταξη και την κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αυτισμό και η συγκεκριμένη ερώτησή μου είναι η εξή. Έχετε στοιχεία που να αναλύουν τις διαφορές αυτές μεταξύ των κρατών μελών και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτές τις σημαντικές αποκλήσεις της εργασιακής ένταξης. Υπάρχουν κοινέ πτυχές και το γνωρίζουμε. Οι επενδύσεις στην παιδεία που αναφέρατε. Ένα συγκεκριμένο και πλήρες νομοθετικό πλαίσιο υποστήριξης των ανθρώπων με αυτισμό. Αλλά έχετε στοιχεία που να συσχετίζουν αναχώρα, ανακράτος μέλος, αυτούς τους παράγοντες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την καλύτερη εργασιακή ένταξη θα μπορούσαμε δηλαδή ως Ένωση να αναπτύξουμε ένα κοινό πλαίσιο. Επίσης, υπόθηκε ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ομάδες ανθρώπων με συγκεκριμένες αναπηρίες, αλλά ακριβώς για το λόγο αυτό πρέπει να αναλύσουμε τις ιδιαιτερότητες, τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε μίας ομάδας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πισλάρου. Θα μιλήσω ρουμανικά, πρόεδρε. Σε σχέση λοιπόν με το θέμα του αυτισμού. Ε, θα έλεγα ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερο θέμα. Εμείς έχουμε ένα οικογενειακό μέλος ε, που χάσαμε από επιληψία στα νεαρά του χρόνια, στην νεότητά του, ακριβώς τη στιγμή που προσπαθούσε να βρει μια θέση εργασίας. Εμείς λοιπόν βιώσαμε το πρόβλημα αυτό κυρίως ως πρόβλημα πρόσβασης και θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ως εξής. Αφενός υπάρχουν διακρίσεις, δυστυχώς, δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ανθρώπων με συγκεκριμένες αναπηρίες όπως ο αυτισμός. Παραβιάζονται λοιπόν τα δικαιώματά τους και υφίστανται οι άνθρωποι αυτοί οι διακρίσεις. Πολύ συχνά η άγνοια είναι αυτή που εξωθεί αυτές τις διακρίσεις δεν δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Και ταυτόχρονα δεν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους. Αλλά θα ήθελα σήμερα περισσότερο να επιμείνω σε μια άλλη πτυχή. Σχετικά με την αρμοδιότητά μας ακριβώς ως Επιτροπή Απασχόλησης. Για την δυνατότητα της κοινωνίας να εντάξει ανθρώπους με αναπηρίες και ανθρώπους κυρίως με αυτισμό. Δεν πρόκειται για δαπάνες, για κονδύλια που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε από το αίσθημα ελέους ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσαμε να, ε, να ε, θεωρούμε συναισθηματικά. Έχουμε, οφείλουμε στο σύστημα της παιδείας μας, οφείλουμε στο κοινωνικό μας σύστημα, να εντάξουμε την ομάδα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τέτοιες αναπηρίες. Οφείλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να βρουν απασχόληση στην κοινωνία μας. Η μεγαλύτερη δυσκολία που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι ότι σημαντικό τμήμα της κοινωνίας ε, τονίζει μόνο τα δικαιώματα. Αλλά καλό είναι αυτό, αλλά χάνουμε την οπτική μας άλλα στοιχεία. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε συγκεκριμένα εργαλεία επενδύσεων. Έχουμε το InvestEU, έχουμε διάφορα πλαίσια ευκαιρίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε να κινητοποιήσουμε προγράμματα υπό την Τράπεζα Επενδύσεων, ώστε να έχουμε καλύτερες συνθήκες σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλους τους εργοδότες που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια ένταξης των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία. και θα ήταν ζωηρή μου επιθυμία κατά τη διάρκεια αυτής εδώ της εντολής, αυτής εδώ της θητείας να μπορέσουμε απτά να συνεισφέρουμε στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη και να μην μιλούμε πλέον για διακρίσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, λέει ο κύριος Μαγιορίνο για την ευκαιρία αυτή, για την συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε την ε, φιλοξενούμενη για την παρουσίαση. Μιλώντας για τον αυτισμό, μιλούμε για πράγματα, για συνθήκες ζωής πολύ διαφορετικές. Αλλά θα έπρεπε σε αυτό το βήμα να αναρωτηθούμε τι μπορούμε στην πράξη να κάνουμε. Και επομένως περισσότερο από ερώτηση είναι μια ιδέα αυτή που σας λέω, μια σκέψη. Θα μπορούσαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Συχνά στην Επιτροπή μας συζητούμε, για παράδειγμα, τον ελάχιστο μισθό. Και προσπαθούμε σε διαφορετικά δημοσιονομικά πλαίσια να δούμε τις μισθολογικές συνθήκες των εργαζομένων στην Ευρώπη για να αποφύγουμε μη αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Αντιστοίχως, Μιλώντας για τις αναπηρίες, επί τη βάση του απολύτως απαραίτητου εκείνου εγγράφου που είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, επί τη βάση του πολύτιμου αυτού εγγράφου, πρέπει να βρούμε, αν θέλετε, επίπεδα εγγύησης αξιοπρεπούς ενημέρωσης και πολιτικών για την ένταξη την κοινωνική και την επαγγελματική των ανθρώπων με αναπηρίες. Εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να είναι ο ρόλος ο δικός μας. Δηλαδή να εγκαταστήσουμε ένα ελάχιστο όριο κάτω του οποίου να απαγορεύεται απολύτως να πάμε ή να βρισκόμαστε. Και ολοκληρώνω, Πρόεδρε, συνθήκες ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες νομίζω σε διάφορες χώρες βεβαίως είναι διαφορετικό το πρόβλημα δεν καλύπτεται επαρκώς από τα διάφορα εθνικά πολιτικά επίπεδα πολλές από τις χώρες μας και περιφέρειές μας είναι σε μεγάλη υστέρηση εδώ μεγάλη υστέρηση και πρέπει λοιπόν ξαναλέω να θέσουμε ένα όριο, ένα κάτω όριο Η κυρία Ραφάλσκα λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εμπειρογνώμανά μας να την ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή της θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια από μένα. Κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε μέχρι τώρα στη συζήτηση, καθότι μιλούμε για ανθρώπους με αυτισμό στην αγορά εργασίας, νομίζω η έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη ίσως, αγωγή, είναι σημαντικό εδώ. Και η φροντίδα που πρέπει να παρέχεται στους ανθρώπους αυτούς πρέπει να αναγνωρίσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους και τις δυνατότητες τους ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε πιο αποτελεσματικά βήματα. Ο συνάδελφος από την Πολωνία αναφέρθηκε σε αυτήν την παγίδα επιδομάτων σχετικά με την απασχολησιμότητα των ανθρώπων με αυτισμό. Αυτό είναι επίσης πιστεύω σημαντικό να το διατηρούμε υπόψη. Ακούσαμε επίσης για τεράστιες αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών, για την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Αυτό απορρέει εκ του γεγονότος ότι έχουμε και τελείως διαφορετικές ιεραρχήσεις κοινωνικών προβλημάτων και τελείως διαφορετικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης τους. Πάντως το φαινόμενο αυτό, το πρόβλημα αυτό γίνεται όλο και οξύτερο και θα πρέπει να εξεύρωμε καλές πρακτικές αντιμετώπισης, επίλυσης του προβλήματος αυτού. Η εμπειρογνώμονας ε, αναφέρθηκε σε πιλωτικά προγράμματα και εξ όσων εγώ κατανοώ στοχεύουμε στη δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων απασχόλησης συνολικά. Η ερώτησή μου είναι από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα πόσοι άνθρωποι έχουν υποφεληθεί. Μπορούμε να ελπίζουμε να έχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει η κυρία Ζαλεύσκα να ευχαριστήσω και την φιλοξενούμενή μας από την Autism Europe. Πιστεύω ότι αυτό που πρέπει εδώ να αναλάβουμε ως δέσμευση είναι ότι θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά στα επόμενα χρόνια όχι μόνο θα εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καλές συστάσεις και συμβουλές, αλλά θα τις υλοποιήσουμε. Επομένως η πρώτη ερώτησή μου προς εσάς είναι δεν θα έπρεπε μήπως να έχουμε μια συζήτηση με όλες εκείνες τις ενώσεις που εκπροσωπούν ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες και λέω ιδιαίτερες ανάγκες και όχι αναπηρίες γιατί στην Πολωνία έχουμε υιοθετήσει νέα ορολογία και αναφερόμαστε έτσι και για τα σχολικά προβλήματα, τα προβλήματα των παιδιών της σχολικής ηλικίας, ειδικέ ανάγκες και στην παιδεία και στην εκπαίδευση. Έχουμε πολύ καλές συστάσεις και προγράμματα και έρευνες που μας δείχνουν ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες πρέπει να έχει κανείς μια εξειδικευμένη προσέγγιση για τα παιδιά, πρέπει να σχεδιάζει, να αναπτύσσει ιδιαίτερους χώρους, όπως αυτούς που αναφερθήκαμε για τους ανθρώπους με, με αυτισμό. Πρέπει να έχει κανείς ειδικά σχολικά βιβλία και εγχειρίδια. Και πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη επίγνωση και γνώση ευρύτερα του πληθυσμού σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Δεν νομίζω ότι οι εργοδότες ε, ε, επιθυμούν να ε, αποκλείουν τους ανθρώπους αυτούς από την αγορά. Πιστεύω ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και γνώσης. Πρέπει λοιπόν να ενημερώνουμε καλύτερα, να συνεργαζόμαστε καλύτερα, να δείχνουμε τι αποτελέσματα έχουμε, γιατί όλα αυτά δείχνουν ότι αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες. Και δεν υπάρχει καμία συμβουλή που μπορεί να στέκει από μόνη μας. Αυτό μας είπε και η φιλεξενούμενή μας. Χρειάζεται εξειδικευμένη προσέγγιση. Για όλες τις ομάδες του πληθυσμού και βεβαίως για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Όλα αυτά έχουν κόστος. Εμείς έχουμε 200.000 παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και ε, δεσμεύσαμε 800 εκατομμύρια σλότη ακριβώς για την ομάδα των παιδιών αυτών κονδύλι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύτως τίποτε άλλο. Επομένως με τέτοιου είδους καλά παραδείγματα μπορούμε να προχωρήσουμε και σε υλοποίηση, εφαρμογή, απτή εφαρμογή. Ο κύριος Φουρλάς. κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εμπειρογνώμονα για την εντελεχή ανάλυση. Ε, Ω νέο Ευρωβουλευτή, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι συνεδριάζουμε στην παρουσία του Επιτρόπου, του κ. Σμιθ, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθουμε ότι είναι εδώ και μα ακούει. Στην πατρίδα μου, πριν από 50 χρόνια, ε, στην Κύπρο, ε, ο αυτισμό ήταν συνώνυμο με την νοητική νηστέρηση. Τόσο πολύ πίσω. Τα άτομα αυτά δεν ήξερε κανένα πώ θα αντιμετωπιστούν. 50 χρόνια μετά θα πω ότι τα άτομα με αυτισμό είναι στις τάξεις των σχολείων από το δημοτικό μέχρι και το γυμνάσιο με συνοδούς τους συμμαθητές τους, οι οποίοι είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση και είναι εκεί για να βοηθήσουν όταν και εφόσον χρειαστεί. Θα σταθώ σε κάτι που υπόθηκε την ευαισθητοποίηση και το πώς ενημερώνουμε. Θα πω ότι και 10 ώρες να μιλάμε εδώ σήμερα μπορεί να μην λάβουμε όσα λάβαμε από το μικρό φιλμάκι που είδαμε ε, που μα έφερε η αγαπητή φίλη. Άρα νομίζω εκεί πρέπει να στραφούμε. Ένα μικρό φιλμάκι του ενό λεπτού εξήγησε σε πάρα πολλού από εμά τι είναι ο αυτισμό, τι είναι το πρόβλημα στην εργασία. Μήπω θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε αξιοποιώντα αυτήν τη λογική. Μικρά βίντεο, ε, μικρέ παρεμβάσει που μπορούν να δείξουν στον κόσμο τι είναι ο αυτισμό. Να έρθει ε, να γίνει κοινωνό αυτού του θέματος νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ αν στραφούν προ αυτήν την κατεύθυνση. Ευαισθητοποίηση με συγκεκριμένο ε, τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με άλλε ε, δύο ερωτήσεις, ε, ο κύριο Σαλίβα πρώτα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προσκεκλημένους μας. Ε, έκαναν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση ε, και μας βοήθησαν να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να εντάξουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, στην αγορά εργασίας. Όσον αφορά όμως τον αυτισμό, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε 7 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση και νομίζω για να τους ε, βοηθήσουμε ε, το κλειδί ε, που υπάρχει και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Αθρών. Το κλειδί είναι λοιπόν είναι εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ε, εκπαίδευση που δεν αποκλεί αυτούς τους ανθρώπους. Αν δεν έχουμε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ε, και αν δεν εκπαιδεύσουμε και τους εργοδότες έτσι ώστε να μπορούν και αυτοί να αναγνωρίζουν τις ε, καθημερινές ε, δυσκολίες, τότε νομίζω δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι αυτοί, ε, τα προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας. Και νομίζω δεν πρέπει να συνεχίσουμε να χάνουμε ανθρώπινο δυναμικό από την αγορά εργασίας, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να ε, βοηθήσουν στην αγορά εργασίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας σε ένα πρόγραμμα δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε, όπως σας είπα, στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που εντάσσονται στο αυτιστικό φάσμα αλλά και για να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους επαγγελματίες, τους εργοδότες με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί η πραγματικότητα των ανθρώπων που εντάσσονται στο αυτιστικό φάσμα. Η κυρία Βέντ, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Θα συνεχίσω στα δανέζικα. Έχουμε λοιπόν οδηγίες ε, που αναφέρουν ότι δεν επιτρέπεται διακριτική μεταχείριση. Αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει, συμβαίνει συνεχώς. Ε, και γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί οι εταιρείες ε, δεν απασχολούν άτομα του αυτιστικού φάσματος ή με ειδικέ ανάγκες. Ε, διότι οι εταιρείε πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα και δεν έχουν ε, χρόνο να αφιερώσουν, είναι πολύ απασχολημένες. Αν όμως είναι κανείς πάρα πολύ απασχολημένος και δεν έχει χρόνο, υπάρχουν ε, πολλοί στη δουλειά που δεν δουλεύουν καλά, με αυτούς θα έπρεπε να ασχοληθούν. Ίσως λοιπόν χρειαζόμαστε πρότυπα εταιρείες ε, στην Ευρώπη που έχουν εισπράξει το μήνυμα, που απασχολούν άτομα του αυτιστικού φάσματος και ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν και όλοι αυτοί ε, μπορούν να παρουσιάσουν τις επιτυχημένες ιστορίες εταιρείε που αποφάσισαν να απασχολήσουν άτομα του αυτιστικού φάσματος γιατί είναι πολύ καλοί, γιατί έχουν τα προσόντα, γιατί έχουν ε, την εκπαίδευση, όχι δηλαδή εταιρείε που θα κάνουν επίδειξη ότι να εμεί απασχολούμε τόσου πολλούς του αυτιστικού φάσματος, όχι, να δείξουν οι εταιρείε ότι απασχολούν άτομα του αυτιστικού φάσματος γιατί είναι ικανά, αποτελεσματικά Βεβαίω ε, και θα πρέπει να ομιλούμε και για τον ε, κατώτατο μισθό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ε, είναι αποτελεσματικοί και θα πρέπει να αμείβονται με βάση τη δουλειά τους. Εάν οι νέοι με του αυτιστικού φάσματος δεν έχουν κάποια προοπτική και δεν υπάρχουν άλλα μοντέλα, τότε και αυτοί γιατί να εκπαιδευτούν. Άρα δηλαδή χρειαζόμαστε πρότυπα ε, ανθρώπων που είναι του αυτιστικού φάσματος, κάνουν καλή δουλειά, ενδιαφέρουσα δουλειά. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε, να δημιουργήσουμε πρότυπα για τους νέους και για τις εταιρείες. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τις καλύτερες πρακτικές ε, στα κράτη-μέλη και έχουμε και καλές πρακτικές ε, από κάποιες μεγάλες εταιρείες που ήδη απασχολούν ανθρώπους με αυτιστικά σύνδρομα, κυρίως με το σύνδρομο Asperger από όσο ξέρω. Εταιρείες της Silicon Valley που είναι ε, πολύ γνωστές μάλιστα, είναι γνωστές ότι ακολουθούν αυτή την πολιτική και δίνουν την ευκαιρία στους αυτιστικούς ανθρώπους. Αυτό είναι σπουδαίο ε, για μας. Πρέπει να ανταλλάξουμε τις καλύτερες πρακτικές και να αρχίσουμε και να παρακολουθούμε και να τις ακολουθούμε. Αυτό είναι ο βασικός στόχος νομίζω και το βασικό πρόβλημα σε κάποια κράτη-μέλη, ότι δηλαδή ε, αρνούνται παρά τα στοιχεία που έχουμε το γεγονός ότι ένας ε, εργοδότης που δίνει δουλειά σε έναν ε, άνθρωπο με σύνδρομο Άσπεργκερ μάλλον θα κερδίσει παρά θα χάσει. Ε, αυτή είναι λοιπόν η κεντρική σταοχή όσον αφορά τις πολιτικές για τους αυτούς ανθρώπους σε όλα τα κράτη-μέλη και σημαντικό είναι να έχουμε τα νέα, να έχουμε πολύ γρήγορα βοήθεια από, μια, από την αιρή ηλικία δεύτερον κοινωνικές υπηρεσίες όχι στους ανθρώπους μόνο που ήδη υπάσχουν, αλλά και στις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Τρίτον, ε, ε, ε, μάλλον, θεραπεία συμπεριφοράς που λειτουργεί ειδικά όσον αφορά τα μικρά παιδιά με αυτισμό σε ορισμένα κράτη-μέλη. Όπως στη Σλοβακία δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτή τη θεραπεία. Οι οικογένειες πρέπει να την πληρώνουν. Οι ίδιες είναι πάρα πολύ δαπανεροί, πάρα πολύ ακριβοί. Δεν μπορούν πολύ συχνά. Και άρα τα παιδιά τους δεν έχουν καμία απολύτως βοήθεια. Τέταρτον βεβαίως είναι η παιδεία που πάει χέρι-χέρι με την κοινωνική ένταξη. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνική ένταξη χωρίς να έχουμε πρόσβαση σε φυσιολογική ε, ε, ποιοτική παιδεία εκπαίδευση για ε, τα παιδιά με σύνδρομο και έπειτα και οι υπηρεσίε έβρεση εργασία πρέπει να αρχίσουν να το λαμβάνουν υπόψη, γιατί μόνο όταν υπάρχουν τέτοιου είδου λειτουργικέ ε, ε, ε, υπηρεσίε θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειέ του, αλλά και οι υπάλληλοι του, γιατί πρέπει εμεί να του μπορέσουμε να του εκπαιδεύσουμε να τους καταρτήσουμε να δουλεύουν με ανθρώπους με ε, προβλήματα. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην καλεσμένη μας για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας, για τις οποίες και σας ευχαριστώ. Γιατί δείχνουν ότι υπάρχει πραγματικό και ειλικρινέ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ όλους, ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής για το feedback, τις προτάσεις σας. Ε, ε, είπατε πολύ σωστά ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια σφαιρική προσέγγιση όταν μιλάμε για αυτισμό. Δεν πρόκειται μόνο για την απασχόληση, πρόκειται για την έγκαιρη παρέμβαση, την πρόσβαση στις θεραπεία και στην παιδεία με τη σωστή στήριξη όμως και συνοδεία. Γιατί αν βάλεις ένα παιδί σε ένα ε, σχολείο ε, γυμνάσιο χωρίς στήριξη θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Πείτε να δούμε και πώς θα αλλάξουμε ε, την εικόνα της κοινωνίας για τον αυτισμό, να ενημερωθεί ο κόσμος, να φτιαχτεί κατανόηση. Ε, πολύ καλή ιδέα ε, είναι το role model που είπατε και την επόμενη, του χρόνου έχουμε μια εκστρατεία ενημέρωσης και σας καλούμε να στηρίξετε την πρωτοβουλία μας αυτή, θα είμαστε σε επαφή. Κάποιος ε, ανέφερε ότι είναι κρίσιμη η, ε, ε, ο χρόνος μετάβασης και πρέπει αυτό να είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μην εγκαταλείπουν επειδή, ανακαλύπτουν, επειδή αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολη κατάσταση, να ανταλλάξουμε καλύτερες πρακτικές, να τοπίσουμε τα καλύτερα πρότυπα στην Ευρώπη. Ξέρουμε κάποιες χώρες που είναι πιο προηγμένες, όπως οι σκανδιναβικές, όπου υπάρχει ειδική φροντίδα, αλλά ούτε καν εκεί δεν είναι όλα τέλεια. συνεχίζουν και εκεί να αγωνίζονται. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια μαγική λύση. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ερευνούμε επίσης για τα τι καταφέρνουν οι άνθρωποι αυτοί και τι προγράμματα τους βοηθούν καλύτερα. Και αυτό είναι πολύ βασικό τομέα. Πρέπει λοιπόν να ε, στηριχθούν οι έρευνες και τα απορίσματα των ερευνών αυτών να διαδίδονται έχουμε, ε, συμμετέχουμε στο ευρύτερο κίνημα ε, για τη, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες. Είμαστε ισχυρότεροι όταν είμαστε ενωμένοι. Κάποιε από τις βασικές συστάσεις είναι συστάσεις που στηρίζει γενικότερα το κίνημα των ε, αναπήρων, ειδικά όταν πρόκειται για τις επόμενες στρατηγικές δηλαδή αναπηρία για, την, για τα άτομα μάλλον με ειδικές ανάγκες. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, αλλά ε, εμείς ε, να σας δηλώσω ότι είμαστε ευτυχείς ε, να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τους ευρωβουλευτές. να σας πω ότι πολύ χαιρόμαστε που στηρίζετε την πρωτοβουλία μας και πόσο ικανοποιημένοι είμαστε που μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Προφανώς το θέμα αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για την Επιτροπή ΕΜΠΛ. Ήταν η πρώτη μας συνεδρίαση, αλλά δεν θα είναι η τελευταία και πιστεύω επίσης πως το θέμα αυτό είναι, ε, αξίζει να συζητηθεί περαιτέρω στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. And the last presentation would be the presentation by the Commission. Uh, commission Τώρα έχουμε την κατεξοδότηση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατεξοδότηση κανονισμού για τη συμπλήρωση κανονισμού κτλ. όσον αφορά τον ορισμό του παπημένων κλιμάκων μοναδίου κόστους των καταπικοπήν ποσών για την επιστροφή δαπανών από την Επιτροπή στα κράτη-μέλη. Καλώς ήρθατε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ανδριάννα Σοκοβά που θα είναι εκείνη που θα μας εξηγήσει ε, τι, περί τίνος πρόκειται. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές. Καταρχάς είμαι εδώ για να σας ε, παρουσιάσω την 8η τροποποίηση του, του, του κανονισμού που υιοθετήθηκε το 2015 αρχικά και θα σας δώσω τον μηχανισμό για τις απλοποιημένες, ε, ε, τον απλοποιημένο υπολογισμό ε, του μοναδίου κόστου που είμαστε, πόσα κρατημέλη, πόσες θεωρήσεις και εποπτήσεις έχουμε κάνει και τι καλύπτει αυτή η 8 τροποποίηση. Ε, ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του 2013 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει κατεξοδότηση κανονισμό ή κατεξοδότηση πράξη για τα, τις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους για συγκεκριμένες συναλλαγές, η δυνατότητα υιοθέτηση ε, των κατεξιδότηση ε, κανονισμών και πράξεων επιτρέπει στα κράτη-μέλη και στους δικαιούχους να έχουν νομική σταθερότητα και ασφάλεια. Οι εθνικοί πάλι γνωρίζουν τι συμβαίνει ακριβώς γιατί όλα αυτά δημοσιεύονται και οι λογιστικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται εθνικά μπορούν επίσης να ε, χρησιμοποιηθούν γιατί αυτό εδώ το σύστημα αφορά μόνο την αποζημίωση, την επιστροφή δαπανών από την Επιτροπή πρόστα προς τα κράτη-μέλη. Οποιαδήποτε διαδικασία λοιπόν και αν έχει χρησιμοποιηθεί αρχικά για να δοθεί κάποια επιχορήγηση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες αυτό δεν εξετάζεται πλέον από τον έλεγχο τη Κομισιόν. Και επίσης σημαντικό είναι ότι όταν όταν αυτές οι διαδικασίες ε, έχουν υιοθετηθεί για συγκεκριμένες ε, συναλλαγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου χωρίς περαιτέρω κοινοποίησης οι διατυπώσει. Το μονοδιαίο <coughs> κόστο ή κατά αποκοπή ποσά που συμπεριλαμβάνονται στην κατεξοδότηση πράξη προτείνονται από τα κράτη-μέλη και έπειτα εμείς κάνουμε μια πολύ λεπτομερή ανάλυση σε διαβούλευση με τι εμπλεκόμενε υπηρεσίε που μπορεί να βοηθήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Εξετάζουμε επί ποιε βάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί και οριστεί αυτέ τι τις κλίμακε κλίμακες μοναδιαίου κόστου, ώστε να αποτελούν ακριβώς αντικατοπτρισμό των μονάδων αυτών που αναφέρονται και έπειτα έχουμε τη δυνατότητα από πλευρά της Κομισιόν να προετοιμάσουμε και να υποβάλουμε με δική μας πρωτοβουλία ένα σύνολο τυποποιημένων κλιμάκων για κάποιες ομάδες ή για όλα τα κράτη-μέλη. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τις δικές μας αναλύσεις και υπολογισμούς γι' αυτό. Υπάρχει εδώ πολιτική δέσμευση και η Κομισιόν θα συνεχίσει να πιέζει, να πιέζει για αυτές τις υποποιημένες κλίμακες γιατί πρώτα απ' όλα Αυτές ε, οι κλίμακες έχουν μεγάλο επιρροή στο ποσοστό σφάλματος ε, ε, και έπειτα η επιστροφή η αποζημίωση βασίζεται στο μοναδιαίο κόστος ή στο ε, καταποκοπικό ποσό. Η τυποποιημένη διαδικασία επιταχύνει την εφαρμογή των προγραμμάτων και επίσης μετακινεί ο κέντρο βάρους από τι χρηματοπιστωτικές δαπάνες στα πραγματικά αποτελέσματα, στην απόδοση των προγραμμάτων. Με αυτόν την 8η ε, τροποποίηση υιοθετούμε τυποποιημένες ε, κλίμακες για 10 επιπλέον κρατημέλη και έχουμε εισάγει εδώ και τις αλλαγές που υιοθετήσαμε πριν από 8 ε, μήνες. Ε, δεν αλλάζει τίποτε άλλο. Ε, έχουμε το ίδιο περιεχόμενο όπως το 2015 επεξηγείται το πεδίο. Μετά έχουμε το, τις τυποποιημένες και στο μοναδιό κόστο, το καταπικοπή ποσό και όπως αυτά ορίζονται στα παραρτήματα ανά κράτος μέλος. Έχουμε ένα παράρτημα για κάθε κράτος μέλος, έχουμε ορισμό των δικτών, της μέτρησης και των ποσών, καθώς και ε, τα κράτη-μέλη ζήτησαν τη δυνατότητα να μπορούν να προσαρμόζονται, ας πούμε, να τα προσαρμόσουν αυτά σε σχέση με τον πληθωρισμό π.χ. Αυτές οι προβλέψεις περιλαμβάνονται στο παράτημα κάθε κράτος μέλους. Ε, πού βρισκόμαστε τώρα. Λοιπόν, βλέπετε ε, τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν με το πράσινο είναι αυτό το χρώμα τέτοιες είδους κλίμακες και η Πορτογαλία θα προσχωρήσει σε εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν αυτή τη, αυτές τις ε, τυποποιημένες κλίμακες του μοναδιαίου κόστους. Ανέφερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ορίζει τέτοιου είδου κλίμακες. Μέχρι τώρα το έχουμε πράξει για την εκπαίδευση, για την εκπαίδευση ανέργων, ε, παροχές ε, συμβουλευτικής και εκπαίδευση απασχολούμενων. Η Πορτογαλία είναι το 28ο κράτος μέλος που θα προσχωρήσει και θα αναφέρω με λεπτομέρειες ποιες χώρες καλύπτονται από αυτόν τον κανονισμό, ποιες είναι οι μορφές κόστους και οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτόν τον κανονισμό. Τροποποιούμε λοιπόν τα παραρτήματα για Τσεχία, Μολδαβία, Ρουμανία, Κύπρος και Ιρλανδία και επίσης ε, θα προσθέσουμε νέα καταποκοπή ποσά για την τεχνική βοήθεια για τη Γαλλία και την Ιρλανδία και Έχουμε ήδη παρουσιάσει αυτή την, ε, τον κατεξιότηση κανονισμό στο Συμβούλιο την 1η Οκτωβρίου. Ο κανονισμός αυτός υιοθετήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μία περίοδος ε, δύο μηνών που δεν πρέπει να κατατεθούν ε, ενστάσεις και το Συμβούλιο μας έχει ενημερώσει ότι σύντομα λύγει αυτή η περίοδος. Η 8η τροπολογία τροπολποιεί επίσης τα παραρτήματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση και αυτό για να υπάρξει προσαρμογή του επίπεδου σε ορισμένα κράτη-μέλη, όπου έχουμε επιτύχει επιπρόσθετες πληροφορίες και έχουμε και ένα παράρτημα που αφορά στην Πορτογαλία. Ας δούμε τώρα ε, ποιες είναι οι λειτουργίες που καλύπτονται ε, για το μοναδίο κόστος μετά την θέσπιση της 8 ε, τροπολογίας. Έχουμε τη Γαλλία, μοναδιαίο κόστος για την που έχει σχέση με μεμονωμένα επαγγέλματα. Ε, επίσης για την επαγγελματική απασχόληση και υπάρχει και πρόσβαση σε περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση. Επιστρέφουμε τις δαπάνες ε, ε, για αυτό το λειτουργικό πρόγραμμα με βάση τον αριθμό των ατόμων που έτυχαν αυτή της απασχόλησης ή απέκτησαν επιπρόστα προσόντα. Υπάρχει επίσης ένα καταποκοπή ποσό για δαπάνες τεχνικής βοήθειας, για προγράμματα που αφορούν ε, τη Γαλλία και το λειτουργικό πρόγραμμα επίσης ε, που αφορά στη Γαλλία. Στην Τσεχία έχουμε 8-9 μοναδιαία κόστη και θέλω να σας πω ότι μέχρι τώρα η Τσεχία έχει 14 τέτοια μοναδία κόστη και ε, στα τρία έχουμε προτείνει τυποποιημένες κλίμακες. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα η Τσεχία θα καλύπτεται από αυτές τις κλίμακες. Άρα δηλαδή είναι σαφές ότι μπορεί να υιοθετηθεί αυτό το μοντέλο επιστροφών ε, και έτσι να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει περισμένο ποσοστό σφάλματος και γρήγορη εφαρμογή. Υπάρχει η τροπολογία για την Μάλτα η οποία ζήτησε αλλαγές σε τέσσερα τέσσερις μορφές ε, μοναδιαίου κόστους. Έχουμε μοναδιαίο κόστος ε, για τις ε, υποτροφίες. Αυτό βεβαίως βασίζεται στα αποτελέσματα. Κατόπιν για την Ιταλία έχουμε εκεί κάποιες εξελίξεις. Μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε άλλα δύο προγράμματα. Ένα εξ αυτών ήταν για τη Λομβαρδία και τους δώσαμε τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν το μοναδιαίο κόστος που έχει ήδη επιβληθεί σε άλλες περιοχές επεκτείνουμε το μοναδιαίο κόστος ε, για τους ε, ερευνητές ε, σε τρεις άλλες περιοχές, Βαλενταώστα, Καμπάνια και Φλωρεντία. Επίσης έχουμε το μοναδιαίο κόστος για την πρωτοβουλία για τους νέους ε, αυτά αφορούν μεμονωμένη εκπαίδευση, γενικότερη εκπαίδευση. Για τη Σλοβακία έχουμε αλλαγές σε πέντε ε, υπάρχοντα μοναδία κόστη. Ε, αυτές οι αλλαγές βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και επίσης καλύπτουμε την Ολλανδία με νέο μοναδία κόστος για την προσφορά επιπρόσθετης ε, εργασίας και κατεύθυνσης. Ε, στη Ρωμανία έχουμε νέο μοναδιακό για την παροχή γευμάτων σε παιδιά ε, και επίσης προβλέπεται ότι θα υπάρξει και προσαρμογή με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Έχουμε μία αλλαγή στο παράρτημα για την Κύπρο. Εκεί έχουμε νέες μορφές μοναδιαίου κόστος για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας Διοίκηση για το λειτουργικό πρόγραμμα απασχόληση ανθρώπινη πόρη και κοινωνική συνοχή. Στην Ιρλανδία έχουμε καταποκοπή ποσό για την τεχνική αρρωγή ε, και επίση έχουμε και ένα νέο μοναδιαίο κόστος για όσους εργάζονται στο πρόγραμμα ΣΥΚΑΠ. Νέο κράτο μέλος είναι η Πορτογαλία, όπως σας είπα, είναι το 28 κράτος που ε, προσχωρεί στον κανονισμό και εκεί προβλέπεται μοναδίο κόστος για ε, άτυπη εκπαίδευση ε, υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Με μεγάλη χαρά έκανα αυτή την παρουσίαση γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ε, τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους. Ε, αυτή τη στιγμή δουλεύουμε σε πέντε κράτη-μέλη για να υπάρξουν νέα τέτοιες ε, τυποποιημένες κλίμακες που σημαίνει ότι ε, το πρώτο εξάμενο του επόμενου έτους θα έχουμε νέα στοιχεία και τα κράτη-μέλη ε, θα μπορούν ε, να ε, επιστρέφουν τις δαπάνες με πολύ πιο απλή διαδικασία. Σας ευχαριστούμε, Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση των τροπολογίων. Παρακαλώ, ο κύριος Πίσλαρο. διαδικαστικά, Πρόεδρε, να ρωτήσω. Αν, πότε κατάλαβα, αν θα έχουμε αντίρρηση από το Συμβούλιο θα είναι απλώς προς ενημέρωσή μας ή μπορούμε να υποβάλλουμε τροπολογίες της ε, κατεξιοδότησης συμπράξης. Και ποια προθεσμία θα έχουμε η διαδικασία αυτή επί του περιεχομένου. Είπατε ότι έγινε μια συζήτηση με πέντε κράτη-μέλη για νέα εκδοχή. Ποια είναι αυτά τα πέντε κράτη-μέλη με τα οποία, εν πάση διαβουλεύεστε κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω και για την παρουσίαση. Εφόσον κατάλαβα καλά, σχετικά με τις ωφέλειες αυτής της απλούστευσης για τα κράτη-μέλη, η Επιτροπή προτίθεται να χρησιμοποιήσει την πράξη αυτή ευρύτερα να καλύψει δηλαδή περισσότερα κράτη-μέλη και περισσότερα είδη λειτουργία ή επιχείρηση, αν κατάλαβα καλά. Αυτό μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο. Δηλαδή ποια είναι τα σχέδια της Επιτροπής ως προς αυτό. Η κυρία Σουκόβα, ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ μιλούμε για κατεξιότητα και 27 Σεπτεμβρίου υφετήθηκε, έχουμε δύο μήνες για τους συνομοθέτες να αποφασίσουν κατά πόσο αποδέχονται ή όχι. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε. Αυτό ισχύει και για το Συμβούλιο προφανώς. Και είναι η πρώτη ε, φορά που δοκιμάζουμε κάτι τέτοιο για εργαλείο πληροφορικής. υπάρχει και η σιωπηρή συνένεση. Δηλαδή, εάν μέχρι τις 27 Νοεμβρίου δεν λάβουμε αντιρρήσει, θα θεωρήσουμε ότι έχετε εγκρίνει. Για τα νέα κράτη-μέλη, Αυστρία και Ρουμανία είναι οι χώρε με τι οποίε είχαμε ενεργό συζήτηση. Δεν μπορώ να θυμηθώ όλες τι χώρε γιατί οι συνάδελφοι που δουλεύουν σε τεχνικό επίπεδο συνεργάζονται με τι αρχέ διαχείριση με την γαμαδελτα budget για να εξασφαλίσουν ότι τα, στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούν είναι ορθά και ασφαλή σχετικά με την απλουστευμένη διαδικασία κόστους και υπολογισμού του. Πάντως έχουμε περισσότερα κράτη-μέλη και δίνουμε λίγο χρόνο και στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν τις δικές τους μεθοδολογίες υπολογισμού. Δεν υιοθετούμε κανονισμό κατεξιότηση για ένα κράτος μέλος όπως αντιλαμβάνεστε. Και νομίζω ότι μπορώ να δηλώσω αισιόδοξη για την απλουστευμένη αυτή μέθοδο. Καταρχάς είμαι 20 μήνες και αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε τα διάφορα επίπεδα απλουστευμένου κόστος που χρησιμοποιούν τα κρατημέλη. Επομένως το μονεδιαίο κόστος το χρησιμοποιούν μόνο για τις αποζημιώσεις τα κρατημέλη. Έχουμε εργαστήρια, σεμινάρια στα κρατημέλη όπου εξηγούμε ότι χρειάζονται περισσότερο. Έχουμε ένα δίκτυο υποστήριξης για την απλούστευση και εκεί συναντώνται όλα τα κρατημέλη που ενδιαφέρονται για τη δικασία απλούστευσης και εκεί συζητούμε ποιες επιλογές σε απλουστευμένο κόστος έχουν απτυχθεί, ποιες δυνατότητες παρέχονται για την ε, ταχεία εφαρμογή των προγραμμάτων και είναι πολύ σημαντικό αυτές οι επιλογές απλουστευμένου υπολογισμού κόστους να μπορούν να προσαρμοστούν αντιστοίχως προς διάφορα κριτήρια ή δείκτες ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Χωρίς πρόσθετους ελέγχους ή άλλες προσαρμογές. Και αυτό είναι αποδεκτό από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε την κυρία Σουκόβα. Να σας θυμίσω το χρονοδιάγραμμα για την Επιτροπή Απασχόλησης. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου. Για το Συμβούλιο ή για το Κοινοβούλιο συνολικά είναι η 27η Νοεμβρίου. Ο κύριος Πίλτσαρο Οπότε διαδικαστικά, Πρόεδρε, εάν μιλούμε για τις 6 Νοεμβρίου, δηλαδή αύριο, επί τη βάση αυτής της παρουσίασης, θα εξετάσουμε το έγγραφο και αν έχουμε σχόλια πώς μπορούμε, λέει ο χωρίς να ολοκληρώσει τη φράση του. Πρόεδρος, αντίρρηση σημαίνει όχι. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Είναι ναι ή όχι. Ναι, Πρόεδρε, το κατάλαβα αυτό. Ήταν απολύτως σαφές και εκτιμώ την παρουσίαση της Επιτροπής. Αλλά ίσως η Επιτροπή θα έπρεπε να έχει έρθει λίγο νωρίτερα εδώ πέρα στο Κοινοβούλιο σε αυτέ τι κατεξιότητε συμπράξει, ώστε στην Επιτροπή Απασχόληση να έχουμε λίγο χρόνο να αποφασίσουμε σε μια αφιερωμένη συνεδρίαση για το κατά πόσον έχουμε αντιρρήσει. Γιατί μου φαίνεται διαδικαστικά ότι δεν θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε καμία. να διατυπώσουμε καμία αντίρρηση. Και δεν είναι ότι έχω αντίρρηση. Διαδικαστικά το λέω. Δηλαδή στο μέλλον. Δεν θα έπρεπε να έρχεται η Επιτροπή λίγο πιο νωρίς ώστε να προλαβαίνουμε να συζητούμε τα θέματα αυτά. Ε, σημείωση από πλευράς μου, λέει η Πρόεδρος. Κάθε μέλος της Επιτροπής έχει ατομικό δικαίωμα να έχει αντίρρηση, δεν εξαρτάται από τους συντονιστές, λέει η Πρόεδρος. Επομένως, αν υπάρχει ατομική αντίρρηση ενός μέλους, πού θα συζητηθεί. Δηλαδή, αν ένα μέλος έχει αντίρρηση, τι θα γίνει τότε. Η κυρία Σούκοβα, λέει ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, λέει ο πρόεδρος, εάν υπάρξει αντίρρηση, θα τεθεί το θέμα στην συνάντηση των συντονιστών. Ο κύριος Πίσλαρου. Εγώ εκτιμώ, πρόεδρε, ότι μας παρουσίασε τον κατεξιότησαν κανονισμό η Επιτροπή και σημαντικό είναι που είμαστε ενήμεροι. Θα ζητούσα από την Επιτροπή την ευγενή καλοσύνη να προσέρχεται λίγο νωρίτερα. να μας παρουσιάζει τέτοια θέματα, γιατί τώρα η διαδικασία είναι αδύνατη, ακόμα και αν υπήρχε επί της ουσίας αντίρρηση από κάποιον που δεν λέω ότι είναι έτσι. Πρόεδρος, η Επιτροπή αυτή κάνει την παρουσίαση επιπροσθέτως προς την γραπτή διαδικασία που είχε λάβει η χώρα νωρίτερα. Μάλιστα, Πρόεδρε, λέει ο κύριος Πίσλαρου, εγώ θα ελέγξω με τους ε, συμβούλους μου να δω τι είχαμε λάβει μέσω email. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Με αυτά ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ευχαριστώ όλους για τα ενδιαφέροντα ερωτήματα και τη βοήθειά σας και την συμμετοχή σας. Τώρα να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 12 του μηνός. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα.